Καλημέρα σε όλους. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα με την ενημέρωση σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών στην συνεδρίαση τη χθεσινή της 6 το απόγευμα. Σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν, οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν γνωμοδότηση και σε, όσα, σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Αλάκη στο συνάδελφο Γκάγερ. Έτσι λοιπόν η γραμματεία θα υποβάλει έκθεση σε σχέση με όσα έγιναν περί Αφγανιστάν στην προηγούμενη θητεία και θα απευθυνθούν και κάποια ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη διαχείριση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονταν και κατευθύνονταν στο Αφγανιστάν. Οι συντονιστές επίσης αποφάσισαν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για τις υποθέσεις που εξέτασε η Όλαφ σε σχέση με το Αφγανιστάν και να μας δώσει συγκριτικά στοιχεία ως προς τις δαπάνες των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών στο Αφγανιστάν. Και αυτό κατόπιν των των πολύ συγκεκριμένων και έντονων δηλώσεων του κ. Αλέκη. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει και μια συνάντηση κλεισμένων των θυρών με την Επιτροπή και την όλα, ως προς το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την αντιπροσωπεία μας στην Ιταλία στις 25 Οκτωβρίου, αποφασίστηκε να γίνουν κάποιες αλλαγές ως προς το πρόγραμμα που αρχικά είχε προγραμματιστεί από τη Γραμματεία ειδικά, ειδικότερα μάλλον, θα προβλέψουμε επίσκεψη για να δούμε πώς υλοποιούνται τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ακούσουμε και τον Γενικό Εισαγγελέα της Ιταλίας, που ασχολείται με θέματα κατά της μαφίας, και ιδίω ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τον καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Για το σημείο Γ, το ερώτημα της Ένωσης ΦΛΕΡ, χρήση δηλαδή του ημικυκλίου του Κοινοβουλίου για την ημερίδα της, ε, κατά της διαφθοράς της 9 Νοεμβρίου και επειδή εκεί μπορεί να συμμετάσχουν τουλάχιστον 500 άτομα ή 700 άτομα, εδώ θα υποβληθεί το αίτημα προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Βούζεκ, ώστε να δούμε κατά πόσο νεύσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για θεσμικές ε, συναντήσεις. Και ω προ τα διάφορα, ζητάτε από τη Γραμματεία να συμφωνήσει με τη Γραμματεία τη Επιτροπή Προπολογισμών ώστε να κανονίσουν μια ημερομηνία για να εξεταστούν οι τροπολογίε του φακέλου για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Έτσι ώστε να ακούσουμε και τον εισηγητή και να μπορέσει να πληρώσει το καθήκον του κατά τρόπο αρμονικό. Επίσης ζητάτε οι συγητές της έκθεσης για το Αφγανιστάν μέσω της ε, διαβούλευσης να ζητήσουν την αποστολή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, κ. Σεύκοβιτς, και υπευθύνου για τις διαθεσμικές και διοικητικές σχέσεις, να ασχοληθεί με το staff screening και τον κώδικα συμπεριφοράς των ανθρώπων. Αυτός προς τη συνάντηση των συντονιστών ε, χθε το βράδυ. Τώρα περνάμε στο σημερινό ραντεβού, το σημαντικό μας ραντεβού, την ακρόαση για τη διαφάνεια στα τυρφωτικά ταμεία, αποδέκτες και δικαιούχοι. Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα προσφυλέ στην Επιτροπή μας βεβαίως του ελέγχου προπολογισμών. Και ήδη από την αρχή της θητείας μας εδώ και ένα χρόνο, ασχοληθήκαμε με ιδιαίτερη αφοσίωση με το θέμα της αφοσίωσης, της, συγγνώμη, ε, διαφάνειας στα διευθυντικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το στοιχείο αυτό είναι καθοριστική σημασία για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την καταπολέμηση της ε, υψηλής ανεργίας που ακόμη συναντάται παντού στην Ευρώπη. Όλα αυτά εξελίσσονται παράλληλα με την πολιτική μηδενική ανοχής ω προς την απάτη, μηδενικής ανοχής ω προς τη διαφθορά και αποφυγής της διασπάθηση των δημοσίων κονδυλίων και πόρων. Δεν θέλουμε να δώσουμε στο οργανωμένο έγκλημα τη δυνατότητα να πάρει στα χέρια του αυτά τα κονδύλια και να ρυπάνει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, την ίδια την πηγή των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, τα διαφορετικά ταμεία. Έτσι λοιπόν έχουμε οργανώσει αυτή τη συνάντηση και ορίζουμε τους προσκεκλισμένους μας, τον κύριο Έρελ Ντέβανη, τον κύριο Τζέρι Μπρίτο. Έρχονται από την Washington, βρήκαν το χρόνο να μας παρουσιάσουν τη δράση μιας ε, σημαντικής χώρας σε αυτό το ιδιαίτερο θέμα. Θα δούμε πώς οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, καλύπτουν το θέμα της διαφάνειας στα δημόσια ταμεία και εδώ μιλάμε πραγματικά για τεράστιους αριθμούς ε, που αφορούν άμεσα τους φορολογουμένους. Και χθε μιλήσαμε για το ξύτατο πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη, που είναι η έλλειψη ενδιαφέροντο των Ευρωπαίων πολιτών ε, προ του ευρωπαϊκού θεσμού. Αυτό κάποιε φορέ οφείλεται και στην έλλειψη διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων κονδυλίων. Καλωσορίζω επίση την κυρία Πελεγκρίν του Κέντρο Βιομηχανικών Σπουδών του Μιλάνου, την κυρία Καταρίνα Ματερνόβα, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια για την Ανάπτυξη, τον Συντονισμό και την Κοινοποίηση τη Πολιτική Συνοχή τη Γενική Διεύθυνση Ρέντιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τον κύριο Λέμπισον, που είναι μέλο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, όπω και τα άλλα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου που ήδη έχουν συνεισφέρει στην Επιτροπή μα, κάνουν εξαιρετικό έργο, πολύτιμο, για τη δική μας για τις δικές μας αρμοδιότητες και για τη σωστή επαλήθευση του πώς δαπανώνται τα δημόσια κονδύλια. Το πρόγραμμα τώρα σύντομα θα έχουμε μια εισαγωγή από τον εισηγητή μας, τον κύριο Λιμπεράτσκι, ο οποίος θα κάνει μια παρουσίαση για την ημερίδα μας. Έπειτα θα δώσουμε το λόγο στους δύο μιλητές που θα μιλήσουν ο καθένας περίπου 20 λεπτά και μετά από αυτές τις δύο παρεμβάσεις θα έχουμε περίπου 30 λεπτά με ερωτήσεις προς τους ομιλητές για ανταλλαγή απόψεων. Και έπειτα θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Και εκεί θα έχουμε συζήτηση που ελπίζω να είναι γόνιμη. Τώρα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Λιμπεράσχη, ο οποίος είναι συγκητής αυτής της πολύ σημαντικής νομοδότησης διαφάνεια στα διευθυντικά από δέκτες και δικαιούχοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω από το εξή: Στη σημερινή οικονομική συγκυρία κάθε λεπτό του ευρώ και κάθε σέντ μετράει και ε, από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Εξού και η συζήτηση για τη διαφάνεια. Η συζήτηση για τη διαφάνεια δεν είναι καινοφανής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 έχει ξεκινήσει την πρωτοβουλία της για τη διαφάνεια. Αλλά όπως συμβαίνει με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, η συζήτηση είχε ξεκινήσει από το παρελθόν, πολύ πιο πριν. Και μία από τις συνιστώσεις είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα περιφερειακά, τα διαστατικά ταμεία για την οικονομική ανάπτυξη παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μιλήσουν και άλλοι αυτό το θέμα και η κυρία Περεγκρίν φαντάζομαι ε, για τη δημόσια διοίκηση, για τη διαφάνεια και τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν επίσης οι πόροι για καλύτερες επενδύσεις και ανάπτυξη και ε, προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης καλούνται να ε, στήσουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου έτσι ώστε να γίνονται σωστά οι δαπάνες. Ωστόσο, όσο καλά και αν είναι τα πρότυπα, δεν λειτουργούν εάν δεν καταλάβουν οι πολίτες και αν δεν βλέπουν οι πολίτες τι γίνεται η ενημέρωση για τη χρήση και τις δαπάνες βοηθάει στην υποστήριξη των πολιτών γιατί γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα χρήματα και έτσι συμμετέχουν περισσότερο στις διαβουλεύσεις για τις μελλοντικές ε, δαπάνες στα διορθωτικά ταμεία. Θα πρέπει λοιπόν να είναι οι μερικοί πολίτες και ε, οι ηθήνονται στα θεσμικά όργανα και μην παραπλανώνται από ε, ψευδή δημοσιεύματα ε, για το πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι. Με 27 κράτη-μέλη και περίπου όλες τόσες γλώσσες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οφείλει να εφαρμόσει τη διαφάνεια με έναν τρόπο πολύ γλωσσικό και πολύ πολιτισμικό. Υποθέτω ότι στι Ηνωμένε Πολιτείε τα πράγματα είναι λιγότερο περίπλοκα από αυτή τη σκοπιά, αλλά είμαι βέβαιος ότι έχουν πολλές άλλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν που αντισταθμίζουν ε, τούτη εδώ. Σήμερα ασχολούμαστε με τα διορθωτικά ταμεία. Αυτό σημαίνει εκατοντάδες δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο η πρωτοβουλία της διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά ε, όλη τη χρηματοδότηση, όχι μόνο τα διαρθωτικά ταμεία. Και θέλουμε να ακούσουμε, κύριε ε, Ντάβανη, για εσά, για τον οργανισμό σας, ε, ανάκτησης, ε, λογοδοσίας και διαφάνειας. Να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημά σας και τι μπορούμε να διδαχθούμε εμείς από εσά. Είναι πρόκληση για μας, λοιπόν, για όλους εμάς, να έχουμε ένα καλό σύστημα διαφάνειας που να μπορεί να εφαρμόζεται παντού στις δημόσιες δαπάνες. Ωστόσο υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα ε, που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και αυτό είναι ότι οι χώρες μας διαφέρουν. Ε, πολλές είναι περιφερειακές, ε, ομοσπονδιακές, έχουν διαφορετικά πρότυπα από κάποιες άλλες ως προς τη διαφάνεια. Και ε, περιμένω να ακούσω την κυρία Πελεγκρίνη γιατί είμαι βέβαιος ότι θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες καθώς και παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής είναι αποτελεσματική και αυτό θα ενισχυθεί πιστεύω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τόσο θα πει η αρμόδια διεύθυνσή της. Επίσης χαίρομαι που θα μας μιλήσει ο κύριος για το ε, τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες ε, και το διαδίκτυο για να έχουν πρόσβαση οι πολίτες. Λοιπόν, περιμένω να μάθω πολλά από σας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να είμαστε υπόλογοι και να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία αυτή οι περισσότεροι πολίτες ε, με το πιο ταχύ τρόπο. Θα ακούσουμε και το ελεκτικό συνέδριο και ήθελα να καλωσορίσω τα εξέχοντα μέλη του Ελεκτρικού Συνεδρίου που είναι σήμερα εδώ παρόντα. Για μας είναι πολύ ευχάριστο αυτό και μεγάλη τιμή. Με τέτοια υψηλή εκπροσώπηση. Να δούμε λοιπόν με ποιον τρόπο ενημερώνουμε τους πολίτες μας. Ως φορολογούμενοι θα πρέπει όλοι να περιμένουμε να είναι γνωστά αυτά τα στοιχεία. Τι υποστηρίζει τι χρηματοδότηση παίρνουν διάφοροι φορείς και διάφορα φυσικά πρόσωπα. Γνωρίζουμε όμως ότι ε, και μια λεπτή ισορροπία εδώ το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων. Ελπίζω η σημερινή ακρόαση να επιτρέψει σε όλους μας να μάθουμε από παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές ε, για θέματα διαφάνεια στη χρήση των δημοσίων πόρων. Και μπορεί να ακούσουμε και για κάποιες δυσκολίες που μας εμποδίζουν να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας. Περιμένω λοιπόν να ακούσω την εμπειρία των ΗΠΑ και προσβλέπω στην ανταλλαγή απόψεων ε, για να βελτιώσουμε τη διαφάνεια που στο κάτω-κάτω είναι ουσιαστικό και αποφασιστικό και για την αξιοπιστία μας και για τη λογοδοσία των διαφόρων οργανισμών μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους εσάς καθώς και όλα τα μέλη της γραμματείας που βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα η σημερινή ακρόαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Λιμπεράτσου. Εδώ πραγματικά αγγίζουμε θέματα ιδιαίτερα ευαίσθητα. Αρκεί να σκεφτούμε ότι σε ό,τι αφορά τα διαφορετικά ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα 2007-2013, μιλάμε για 8.300 ευρώ. Και η Επιτροπή Ανάκτησης και Πανεπένδυσης όπως έχει οργανωθεί από τον κύριο Ομπάμα και που προεδρεύει ο κύριος Ντεβένη, ασχολείται με ποσά του τάξης των 780 εκατομμυρίων δολαρίων. Δις συγγνώμη. Οπότε, μιλάμε για ποσά τεράστια. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε περίπτωση διασπάθησης ή κακοδιαχείρισης. Ένα άλλο σκέλος που αφορά την, το θέμα μας, τη διαφάνεια δηλαδή, είναι και οι δημοσίευση στον ιστότοπο των δραστηριοτήτων των διαφορών επιτροπών, ώστε οι φορολογούμενοι απευθεία να γνωρίζουν ποιε είναι οι ροές των δημοσίων κονδυλίων. Κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντική και η δήλωση αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη εντολή, που έχει αναλάβει, να προάγει την εποπτεία και τον έλεγχο των ε, δημοσίων κονδυλίων για να αποφύγει τη διασπάθηση και την κακοδιαχείριση των κονδύλων αυτών, ώστε να προβάλλονται προς το κοινό όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό επιτρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί και η Επιτροπή αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου προεδρεύει ο κ. Ντέβεν, όπως σας είπα, ορίστηκε τον Φεβρουάριο του 2009 ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, υπεύθυνο να διαχειρίζεται αυτά τα 780 δις ευρώ, να παρακολουθεί τη διαχείρισή τους μάλλον. Επίσης ο Γενικός Επόπτη Γενικός Επόπτης Ίντεν, ο οποίος εργάζεται εσωτερικά στην Επιτροπή αυτή, ανέλαβε σοβαρές δημόσιες έρευνες για θέματα διαφθορα, διαφθοράς, ο οποίος ε, τελικά κατέληξε και στην καταδίκη του κυρίου Αμπράμου στην Washington. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη συμμετοχή σας αυτή την σημαντική ακρόαση για την ε, διαφάνεια και πραγματικά θέλουμε να γνωρίζουμε όλες αυτές τις δράσεις σε σχέση με την παρακολούθηση της διαχείρισης των δημοσίων κονδυλίων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους τους βουλευτές. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα εδώ. Έχω εργαστεί στην κυβέρνηση των ΗΠΑ περίπου 40 χρόνια και είχα πολλές ευκαιρίες να μιλήσω μπροστά στα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Αυτή είναι όμω η πρώτη φορά που επισκέπτομαι το Κοινοβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν τιμή και προνόμιο να μιλώ σήμερα για τα θέματα των διαφανών, τη διαφανού διαχείριση με λογοδοσία. Τα θέματα αυτά είναι δύο θέματα τα οποία με έχουν παθιάσει σε όλη τη διάρκεια τη θητεία μου και τη καριέρα μου. Ιδίω από τότε που ο πρόεδρο Ομπάμα με όρισε ω πρόεδρο τη Επιτροπή Λογοδοσία και Διαφάνεια τον Φεβρουάριο του 2009. Του τελευταίου 17 μήνε, λοιπόν, έχω ζήσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα διαστήματα τη σταδιοδρομία μου. Και θα ήθελα να σα παρουσιάσω τι εμπειρίε μου σήμερα το πρωί. Όπω πολλοί από εσά γνωρίζετε, το Συμβούλιο Λογοδοσία και Διαφάνεια για την ανάκτηση έχει οριστεί βάσει του νόμου για την ανάκτηση και την επανεπένδυση του 2009. Αυτό ήταν μια άμεση απόκριση στην οικονομική κρίση των ΗΠΑ και ο πρόεδρος Ομπάμα υπέγραψε την, το νόμο αυτό τον κύρωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2009. Έχει τρει στόχου ο νόμο αυτό. Να δημιουργήσει νέε θέσει εργασία και να διασώσει τι υπάρχουσες, Να αναθερμάνει την οικονομική δραστηριότητα ώστε να υπάρξουν επενδύσει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να στηρίξει επίπεδα λογοδοσία και διαφάνεια που δεν είχαμε στο παρελθόν για την δημόσια διαχείριση. Υπάρχουν δύο εντολέ για το Συμβούλιο μα εδώ για τον τρίτο στόχο που αφορά τη λογοδοσία και την διαφάνεια η διτή αποστολή μα είναι να ορίσουμε και να διατηρήσουμε έναν ιστότοπο που να είναι φιλικό προ το χρήση και σκοπό έχει να δείχνει στου πολίτε πώ τα δολάρια τη ανάκτηση δαπανώνται και επίση να συντονίζει και να παρακολουθεί τη διαχείριση των 787 δισεκατομμυρίων δολαρίων των ε, ταμείων ανάκτησης, καθώς και να προλαμβάνει την απάτη, την κατασπατάληση ή τις καταχρήσεις. Έχουμε επίσης 10 γενικούς ε, επιθεωρητές που συμμετέχουν σε ένα διοικητικό συμβούλιο και ο Πρόεδρος ε, όρισε εμένα ως Πρόεδρο μαζί με δύο γενικούς επιθεωρητές στο 13 μελές συμβούλιο. Εργαστήκαμε σήμερα με δύο σημαντικές, ε, σύντομα με δύο σημαντικές πρωτοβουλίες και δημιουργήσαμε τον ιστότοπο που είναι γνωστό ως www.recovery.gov έτσι αναλάβαμε και συγκεκριμένε ε, εξουσίε και βάσει του νόμου τη ανάκτηση ω συμβούλιο. Συγκεκριμένα μπορούμε να ελέγχουμε και να υποπτεύουμε τι ε, δαπάνε είτε, ε, είτε με δική μα πρωτοβουλία είτε σε συνεργασία με του ομοσπονδιακού γενικού επιθεωρητέ. Επίση μπορούμε να εκδίδουμε κλητεύσει για να παρακολουθούμε τις ευθύνες και να τις ελέγχουμε, να παραπέμπουμε υποθέσεις απάτης, κατασπατάληση και κακοδιαχείριση τους ομοσπονδιακούς γενικού επιθεωρητές, να διεξάγουμε δημόσιες ακροασει και να καλούμε μάρτυρες και να οργανώνουμε έρευνε, αναλύσει και ελέγχου. Καταλαβαίνω ότι οι παρατηρήσει μου μεταφράζονται ταυτόχρονα σε 15 γλώσσε, οπότε θα ήθελα να σα εξηγήσω λίγο το, τον όρο Γενικό Επιθεωρητή, σε όσου δεν γνωρίζουν καλά τι σημαίνει αυτό. Οι γενικοί ε, επιθεωρητέ είναι ε, οι υπεύθυνοι τη κυβέρνηση τη ΗΠΑ που ασχολούνται με τα θέματα οικονομία και αποτελεσματικότητα, ώστε να ε, εντοπίζουν περιπτώσει απάτη, κατασπατάληση και παραβίαση. Ορίζονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και εγκρίνονται από τη Γερουσία. Οι βασικέ του αρμοδιότητε είναι να διεξάγουν και να παρακολουθούν ελέγχου και έρευνε σχετικά με τα προγράμματα των συγκεκριμένων υπηρεσιών του, να παρέχουν ηγετική καθοδήγηση και συντονισμό και να συστήνουν πολιτικέ για τι δραστηριότητε που έχουν σκοπό να προωθήσουν την οικονομία, την αποτελεσματικότητα και την δραστικότητα στην ε, διαχείριση των κυβερνητικών προγραμμάτων και παραδοσιακά περνούν πάρα πολύ χρόνο ανοιχνεύοντας περιπτώσεις απάτης ή ε, σπατάλης ή εξετάζοντας τέτοιες δραστηριότητες μέσω ελέγχων και ποινικών ερευνών. Τα παραδοσιακά τους εργαλεία είναι καθοριστικά και για την δική μας βασική αποστολή του Συμβουλίου. Και η διατύπωση του νόμου του 2009 εξηγεί ότι οι γενικοί επιθεωρητές θα πρέπει να ασχολούνται με τον περιορισμό του κινδύνου που έχουν να κάνουν ε, με την διανομή και την κατανομή τόσο σημαντικών ποσών χρηματικών, καθώς και τις ε, περιπτώσεις όπου θα μπορούσε να προκύψει απάτη κακοδιαχείριση πριν αυτό συμβεί. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια σημαντική μετατόπιση εδώ. Αυτό η πρόληψη δηλαδή, είναι ένα σημαντικό μέρος της λογοδοσίας της δυτής μας αποστολής. Ε, και η δική μας ε, δράση παρακολούθηση στον τελευταίο 1,5 χρόνο μας έχει οδηγήσει σε πολλές επιτυχίες την πρόληψη απάτης και κοδιαχείρισης ή σπατάλης για τα ομοσπονδιακά κονδύλια. Ένας από μια από τις κλασικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε είναι να εντοπίζουμε τους υψηλού κινδύνου δικαιούχους ε, για τις ομοσπονδιακές συμβάσεις δωρεές και εδώ λοιπόν έχουμε μια διαδικασία σε τρία στάδια. Σε μια πρώτη φάση οι αναλυτές μας στο επιχειρησιακό κέντρο ανάκτησης στην Washington ασχολούνται με την εντοπισμό των συγκεκριμένων δικαιούχων υψηλού κινδύνου. Η διαδικασία screening είναι διαθέσιμη στο κοινό και διασφαλίζει ότι οι ομοσπονδιακοί υπεύθυνοι ε, έρχονται σε συναλλαγές μόνο με εγκεκριμένους φορείς. Για παράδειγμα, εξετάζουμε την οικονομική ιστορία, τον το ποινικό ιστορικό των δικαιούχων, το φορολογικό, τη φορολογική τους κατάσταση. Βλέπουμε αν στο παρελθόν υπήρχε πρόβλημα με κυβερνητικές αρμοδιότητες που είχαν αναλάβει οι φορείς. Και έτσι εντοπίζουμε τον κίνδυνο απάτης. Έπειτα αναπτύσσουμε τα εργαλεία όταν χρειάζεται να αποκαλύψουμε τι μη διαφανεί υψηλού κινδύνου σχέσει μεταξύ φορέων. Έχουμε διάφορα εργαλεία, καθώ και συμμετοχή πολλών επαγγελματιών που έχουν πείρα στο θέμα του ελέγχου, των ερευνών, των προμηθειών, των αναλύσεων προγραμμάτων, τη στατιστική και την εξέταση συνολικών δεδομένων. Έτσι, με τον εντοπισμό των υπόπτων έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Ε, το τρίτο στάδιο είναι να δημιουργήσουμε μοντέλα για να εντοπίσουμε τους παράγοντες κινδύνου και τις σημερινές τάσεις, ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο εργαλείων διαχείρισης για την συνολική μας παρακολούθηση. Για παράδειγμα, δημιουργούμε χάρτες που καθορίζονται οι κομιτείες στο σύνολο των ΗΠΑ και βλέπουμε που έχουν πληγεί περισσότερο από την ύφεση συγκεντρώνουμε δεδομένα για τους δικαιούχους για να εντοπίσουμε τομείς περιοχές κινδύνου και επίσης χρησιμοποιούμε την άμεση γραμμή επικοινωνίας για να μπορούμε να συγκεντρώνουμε στοιχεία για ενδεχόμενα απάτης, κακοδιαχείρισης ή σπατάλης. Και βασιζόμαστε και στην παρακολούθηση της κοινότητας ε, για να εντοπίζουμε τους ανθρωπίνους πόρους όπου ε, χρειάζονται περισσότερο στις Ηνωμένε Πολιτείες, στη χώρα μας. Όλοι λοιπόν οι υπεύθυνοι τη εκπαίδευση και τη ευαισθητοποίηση, καθώ και τα μέλη του Συμβουλίου μα και οι γενικοί επιθεωρητέ σε κάθε κοινότητα, έχουν ε, έρθει σε επαφή με τι ομάδε πολιτών, μέλη του Κογκρέσου, με τα με του υπευθύνου μέσων μαζική ενημέρωση για να γνωστοποιήσουν τι δράσει μα. Επίση, έχουμε πολλέ επιτροπέ, εταιρικέ σχέσει και ομάδε εργασία για να προσπαθήσουμε να φέρουμε αποτελέσματα πριν την απονομή των ε, συμβάσεων των δωρεών και των δανείων. Έτσι λοιπόν, δίνοντα ιδιαίτερε εξουσίε στου γενικού επιθεωρητέ επίπεδο κοινότητα για τη λογοδοσία, αυτό μα μας ε, επιτρέπει να βελτιώσουμε και τον ιστότοπό μα και σε, με μια σχέση συνεργασία να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό εργαλείο στου δύσκολου καιρού που τώρα διανύουμε. Θα ήθελα τώρα να αλλάξω κάπως ε, θέμα και να σας πω ποια, τι πιστεύω για, τις, για τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την διαφάνεια. Ο νόμος της ανάκτησης και της επανεπένδυσης που επιτρέπει τη δημιουργία του Συμβουλίου μας έχει να κάνει με τη χρήση των κονδυλίων, γι' αυτό δημιουργήθηκε αρχικά και ο ιστότοπος που ονομάζεται www.federalreporting.gov για να συλλέγουμε δεδομένα. Εκεί κάθε δικαιούχος των κονδυλίων ε, καταγράφεται, καταγράφεται ως προς τα δεδομένα δαπάνης και μιλάμε εδώ για ένα ιστότοπο που δεν έχει δημόσια πρόσβαση. Εκεί μια ομάδα προγραμματιστών και αναλυτών επεξεργάζεται κάποια δεδομένα που τελικά δημοσιεύονται στον ε, ιστότοπο που είναι ανοιχτό για το κοινό. Επίσης, οι Αμερικανοί μπορούν ε, μέσω της δικής τους κοινότητας και της δικής τους παρακολούθησης να δουν πώς ακριβώς ε, τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από αυτό το νόμο λειτουργούν πώς εξελίσσονται. Μπορούμε, ο μέσο, μπορεί ο μέσος Αμερικανός καθημερινά να παρακολουθεί τις χρηματικές ροές. Και μόλι οι πολίτε μα εντοπίζουν κάτι που πιστεύουν ότι δεν πάει καλά, είναι ελεύθεροι να έρθουν σε επαφή μαζί μα και να το επισημάνουν. Μιλάμε λοιπόν πλέον ε, μεταξύ μα για πολίτε που λειτουργούν ω γενικοί επιθεωρητέ. Καταλαβαίνετε ότι σε όλο τον κόσμο σήμερα διαφάνεια και η λογοδοσία είναι κάτι που ε, ξεπερνάει τα σύνορα των φορέων και των χωρών. Η έννοια της ε, διαφανούς διακυβέρνησης είναι κάτι που έχουμε από την ε, αρχαία Αθήνα όταν οι πολίτες συναντιόνταν στην αγορά για να συζητήσουν τα θέματα της πόλης. Βέβαια, σήμερα έχει περάσει αυτός ο καιρός, ε, οι πληροφορίες και οι ενημέρωση ανταλλάσσονται στο διαδίκτυο και έτσι μαθαίνουμε τα πάντα για τις ε, δράσεις των κυβερνήσεων. Η διαφάνεια λοιπόν είναι ένα τρόπο σε κάθε κυβέρνηση να δίνει στου πολίτε το δικαίωμα να παρακολουθούν την διαδικασία λήψη αποφάσεων. Το να λύνονται προβλήματα, να υπάρχουν καινοτόμε λύσει, να αντιμετωπίζονται προκλήσει και να επιτυγχάνονται στόχοι είναι σημαντικό ε, ω προ το να μπορούν όλοι να παρακολουθούν πώ εξελίσσεται η σχετική διαδικασία. Οι, οι πολιτικοί ηθήνοντε, βέβαια μπορεί κάποιες φορές να μην θέλουν να μοιραστούν τις πληροφορίες, να μην τι να κοινοποιήσουν, αλλά πολλές φορές οφείλουν να το κάνουν. Άλλωστε, ήδη στην αρχή της λειτουργίας του Συμβουλίου μας, ε, στην πρώτη διαδικασία συλλογής εκθέσεων, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν κάποια σφάλματα στην καταγραφή των στοιχείων. Αυτό ήταν ένα μεγάλο δείγμα και ήταν, όπως είδαμε, πολύ πιο εύκολο να το συζητάμε το όλο θέμα της διαφάνειας παρά να το αντιμετωπίζουμε. Όμως, το να αντιμετωπίζουμε την δυσφορία που πολλές φορές προκαλούν τα ασφάλματα που έχουν γίνει στο παρελθόν, τελικά έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα ότι αντιμετωπίζονται τα πράγματα εγκαίρως και διορθώνεται η μη κατάλληλη συμπεριφορά. Τώρα βρισκόμαστε στην τέταρτη περίοδο συλλογή εκθέσεων και πρέπει να πω ότι η ποιότητα και η ακρίβεια των δεδομένων μα έχει βελτιωθεί. Βελτιώνεται με κάθε κύκλο συλλογή εκθέσεων και ελπίζω ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και στι μελλοντικέ περιόδου συλλογή εκθέσεων. Η διαφάνεια, όπω καθορίζεται από του σχεδιαστέ του νόμου του 2009 και τη ανάκτηση, επιτρέπει στου φορολογουμένου να παρακολουθούν καλύτερα την λογοδοσία την κυβερνητική ω τη δαπάνη των ε, ε, δολαρίων που με κόπο έχουν ε, παραχθεί, έχουν, κερδιθεί, έχουν επενδυθεί και έχουν κατανεμηθεί σε δικαιούχος και μπορούν να παρακολουθήσουν σήμερα με τη δική τους κρίση εάν αυτά γίνονται ορθώς, σε συγκεκριμένα μάλιστα προγράμματα. Βέβαια, το να ανταλλάσσονται απλώς στοιχεία για τα δεδομένα δαπανών ε, σε έναν ιστότοπο δεν είναι ο ορισμός ο ίδιος της διαφάνειας σημαίνει ότι με διαφανή μέσα υπάρχουν χρήσιμα δεδομένα τα οποία μπορούν να ενημερώνουν τους πολίτες. Ιδίω σε ό,τι αφορά την διαφάνεια των δαπανών. Τα δεδομένα πρέπει να είναι και επίκαιρα και πρόσφατα και ακριβή και αξιόπιστα. Η δική μου άποψη είναι ότι αν τα δεδομένα προκαλούν σύγχυση στο κοινό, τελικά η διαφάνεια θα δώσει λανθασμένη εντύπωση. Δεν θα γίνει αντιληπτή ω κάτι το θετικό. Πιστεύω πάντω ότι το ίδιο που ισχύει για τη διαφάνεια είναι κάτι που μπορεί να προάγει και την λογοδοσία. Εδώ χρειαζόμαστε σημαντικό λογισμικό και τους ανθρώπινους πόρους μας, αυτά που διαθέτει δηλαδή το Συμβούλιο στο επιχειρησιακό μας κέντρο, ώστε να παρακολουθούμε την κάθε σύμβαση, την κάθε δωρεά και το κάθε δάνειο, για να δούμε πώς ακριβώς έχουν επενδυθεί τα δολάρια και να προβλέψουμε που μπορεί να προκύψουν προβλήματα. Ε, το σύνολο των γενικών επιθεωρητών έχουν βρεθεί σε μια πολύ θετική θέση όσο ποτέ στο παρελθόν και ελπίζω ότι αυτή η, αυτό υποδειγματική, αυτή η λειτουργία θα είναι κάτι που θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ήθελα τώρα να κάνω και δύο τελικές παρατηρήσεις. Ε, το τελευταίο 1,5 χρόνο είδα από προσωπική άποψη πώ η διαφάνεια δίνει εξουσίες στου ίδιου του πολίτε. Με την ψηφιακή επανάσταση σε όλο τον κόσμο βλέπουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αναπόφευκτο να επιδιώκουμε την διαφάνεια. Το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα που έχουν φωτογραφικέ μηχανέ, ε, η παρακολούθηση από τα μέσα μαζική ενημέρωση είναι κάτι που έχει δώσει τη δυνατότητα ενημέρωσης σε όλους τους πολίτες. Νομίζω λοιπόν ότι το στότοπό μας, το www.gov, είναι κάτι που δίνει στους πολίτες την ευκαιρία και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ε, όλη δράση της κυβέρνησης και να την παρακολουθούν εμπιστοποιούμενοι. Και τέλος, νομίζω ότι η διαφάνεια πραγματικά λειτουργεί και από την άλλη πλευρά τη κυβέρνηση και την επηρεάζει. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι αυτή η αρχή έχει οδηγήσει εδώ και τέσσερι δεκαετίε τον τρόπο που λειτουργούν οι δημόσιε υπηρεσίε. Δηλαδή, η διαφάνεια και η λογοδοσία μπορεί να καθορίσει ισοτικό, να ισοτικό ρόλο ω προ το πώ η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα κονδύλια τη. Δηλαδή, καταλαβαίνει <clears throat> ότι έχει να λογοδοτήσει ω προ του συμπολίτε που θέλουν όχι μόνο να βλέπουν, αλλά να πιστεύουν ότι έχουν δικαίωμα να βλέπουν πώ δαπανώνται τα κονδύλια. Έτσι λοιπόν ε, νομίζουμε ότι το Συμβούλιο μας δημιουργώντας αυτό τον ε, ιστότοπο αυτή την πύλη μπορεί να ε, ενημερώσει αποτελεσματικά τους πολίτες για το πώς κροδεύονται τα κονδύλια της κυβέρνησης. Εδώ θα ήθελα τώρα να, παραθέσω και τον James Μάντισον, τον τέταρτο πρόεδρο της χώρας μας, ο οποίος σε μια ομιλία του από τις αρχές του 19ου αιώνα έλεγε κάτι που εδώ και 200 χρόνια παραμένει επίκαιρο, ότι μια δημοφιλής κυβέρνηση χωρίς την κατάλληλη πληροφόρηση δεν μπορεί παρά να είναι μια, ένας πρόλογος για μια κομμωδία ή μια τραγωδία και τα δύο. Σας ευχαριστώ και πάλι που με ακούσατε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για αυτήν την ομιλία, πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας παρουσιάσατε κυβερνητικές λειτουργίες και συμμετοχική βέβαια, τη συμμετοχική διάσταση της κοινωνίας των πολιτών. Τα δημοσία κονδύλια ε, σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν το έθνος, το όφελος και τους πολίτες. Κάποια ιδιωτική τοπίο βέβαια έχουν ανακύψει στις ΗΠΑ, έχουν εμφανιστεί ε, για την παρακολούθηση του πώς δαπανώνται τα δημοσία κονδύλια. Ο κύριος ε, Μπρίτο, ανώτερος ερευνητής του Πανεπιστημίου George Mason της Washington, είναι υπεύθυνο και για το πρόγραμμα πολιτικής ενημέρωσης του ίδιου κέντρου και ασχολείται με τις τεχνολογίες και τις τηλεπικοινωνίε για την πολιτική, με τη διαφάνεια τη κυβερνητική δράση και τη λογοδοσία. Είναι συν ε, του ιστοτόπου για την παρακολούθηση των δράσεων αυτών, ιστότοπος που έχει σκοπό να ενθαρρύνει τους Αμερικανούς πολίτες να ευαισθητοποιηθούν για τα θέματα αυτά και να τα συζητούν ε, σε επίπεδο κοινότητα και πολιτεία. Ήθελα λοιπόν να σα ευχαριστήσω για την παρουσίαση τη πείρα σα αυτή που είναι πολύ χρήσιμη και για το δικό μα το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτή τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, λέγομαι Τζέρι Μπράιτο και είμαι ερευνητή στο κέντρο Μερκάτου του Πανεπιστημίου George Mason τη Βιργινία. Τα τελευταία χρόνια η έρευνά μου βασίστηκε στο πώ οι τεχνολογίε του Ιντερνετ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνηση και του πολίτε για να αυξηθεί η διαφάνεια και να υπάρξει μεγαλύτερη λογοδοσία. Και θα σα αναφέρω ορισμένε από τι σκέψει μου. Η δημοκρατία βασίζεται στην αρχή ότι η εξουσία πηγάζει από τη συνένεση των κυβερνομένων αυτή η συνένεση βέβαια δεν έχει και πολύ νόημα εκτός εάν είναι πληροφορημένος ο πολίτης. Αν η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις μυστικά και αυξάνεται η δωροδοκία και η διαφθορά, τότε η λογοδοσία μειώνεται. Γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στην διακυβέρνηση. Όταν οι επίσημες συνεδριάσεις είναι ανοιχτές στους πολίτες και τον τύπο, όταν τα δημοσιονομικά είναι γνωστά και όταν η νομοθετική διαδικασία είναι ανοιχτή στη συζήτηση, τότε υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία της κυβέρνησης και άρα η διαφάνεια δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά απλώς ένα μέσον προς τον σκοπό που είναι η λογοδοσία. Οι ιδρυτές των ΗΠΑ το αναγνώρισαν αυτό, διότι το Σύνταγμα απαιτεί το Κογκρέσο να κρατά πρακτικά των διαδικασιών του, να καταγράφει τις ψηφοφορίες του και από καιρού καιρό να τα δημοσιεύει όλα αυτά. Και γιατί, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε τι πράττει η κυβέρνηση για να μπορούμε να κρίνουμε την δράση της. Πρέπει να ξέρουμε πώς ψηφίζουν, πώς δαπανούν τα χρήματά μας, ποιον συναντούν και ποιος τους χρηματοδοτεί. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε λογοδοσία και να αποφασίζουμε ποιον να προσλάβουμε και ποιον να διώξουμε. Οι ψηφοφορίες πάντοτε ήταν βέβαια δημόσιες και οι προπολογισμοί το ίδιο, αλλά δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση σε όλα αυτά. Οι σημειώσεις για τις συνεδριάσεις, οι αριθμοί, όλα αυτά για να τα μάθει κανείς πρέπει να πάει σε τίποτε υπόγεια στην Ουάσιγκτον και να τα ψάχνει ολόκληρες μέρες. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ο τύπος για να δείχνει πότε έχει σημειωθεί κάποια παράληψη. Αλλά το ίντερνετ μας δίνει μια, την ευκαιρία να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Η τεχνολογία του ίντερνετ δεν μειώνει μόνο το κόστος της πρόσβασης στην πληροφόρηση, αλλά καθιστά πολύ ευκολότερο για τον πολίτη και το να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει την πληροφόρηση. Με αποτέλεσμα ο καθένας να μπορεί να παίξει ρόλο ρεπόρτερ ή επιθεωρητού. Η διάθεση των πληροφοριών της κυβέρνησης είναι υπέρ του ατομικού χρήστη αλλά επίσης απλοποιεί τη δυνατότητα να συνδυάσει κανείς στοιχεία για τη δράση της κυβέρνησης. Έτσι μπορεί και η ίδια να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Παραδείγματο χάρη, στοιχεία για την ομοσπονδιακές δαπάνες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε ένα τρίτο μέρος όσο χάρτης διαδραστικός που να δείχνει πού πηγαίνουν τα διάφορα κονδύλια. Όσο υπάρχουν τα δεδομένα στο ίντερνετ, τόσο καλύτερα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Ο όρος δομημένη πληροφόρηση είναι κάτι γνωστό. Σημαίνει ότι η πληροφόρηση δίνεται με μορφή εύληπτη, έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα είτε αλφαβητικά είτε ανακεφάλαιο είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιτρέπει μια ιστοσελίδα που δεν είναι στατική. Όταν η κυβέρνηση δίνει τέτοια στοιχεία ανοίγει τον, την πόρτα σε καλύτερη πληροφόρηση στον πολίτη. Υπάρχει και το εργαλείο που ονομάζεται στο ίντερνετ Mashup που δίνει την ευκαιρία στο χρήστη να καταλάβει καλύτερα ποια είναι η δράση της κυβέρνησης. Ο συνδυασμός των στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει νέο τύπο πληροφόρηση. Τα μάσα από αυτά αποτελούν πολύ μεγάλο δυναμικό για τη μελλοντική μορφή που θα πάρει η πληροφόρηση. Αλλά κυρίως δημιουργούν διαφάνεια στην δράση της κυβέρνησης και δείχνουν πόσο σημαντικά μπορεί να είναι ορισμένα δεδομένα που μπορεί να φαίνονταν στην αρχή ασήμαντα. στον ιστότοπο maplight.org φαίνεται τι καλή χρήση μπορεί να γίνει από τέτοια συνδυασμένη χρήση δεδομένων. Γιατί συνδυάζει ας πούμε τις ψηφοφορίες του Κογκρέσου με τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί, τη χρήση των κονδυλίων μάλλον. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτή την τράπεζα δεδομένων του MapLight μπορεί ο χρήστης να δει κάποιο νομοσχέδιο πώς ακριβώς έχει χρησιμοποιηθεί, πού έχει καταλήξει και ποιος τάχθηκε υπέρ και κατά. Επίσης μπορεί να δει πώς ψήφισαν τα μέλη του Κογκρέσου και ποιος χρηματοδότησε τα πάντα. Ποιος ε, έλαβε μέρος στη συζήτηση μάλλον. Αν αυτά τα στοιχεία είναι πάντοτε ανοιχτά και εύληπτα για το χρήστη, μπορεί ο καθένας να καταλάβει ποιες είναι οι διασυνθέσεις που μπορούν να γίνουν, αλλά παρόλα αυτά δεν γίνονται όλα αυτόματα, χρειάζεται η ανθρώπινη κρίση. Χρησιμοποιώ συχνά τον όρο crowdsourcing και εννοώ την μικρή συμβολή ενός ατόμου από ε, μεταξύ εκατομμυρίων για να δημιουργηθεί κάτι που προηγουμένως απαιτούσε να γίνει από ένα άτομο ή μία οργάνωση. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας ε, πω την εμπειρία μου ως πολίτου που δημιούργησε μία τέτοια εφαρμογή crowdsourcing χρησιμοποιώντας στοιχεία από την κυβέρνηση. Και θέλω να σας δείξω ότι αν η κυβέρνηση διαθέσει αυτά τα ασυνδίαστα στοιχεία κάποιος ερευνητής σαν και μένα μπορεί να δημιουργήσει ολόκληρη εφαρμογή που να βελτιώνει την λογοδοσία. Το Δεκέμβριο του 2008 ο Μπαράκ Ομπάμα εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν είχε ακόμη να λάβει τα καθήκοντά του. Παρ' όλα αυτά είχε δηλώσει ότι θα αύξανε τις δαπάνες. Πολλοί είχαν θεωρήσει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να μην διέθετε αρκετά προγράμματα και σχέδια τα οποία να χρησιμοποιήσει για τα κονδύλια που θα τις διατίθενταν. Αυτά τα ονομάσαμε σχέδια έτοιμα για το φιάρι, δηλαδή Shovel Ready Project. Σχέδια δηλαδή που θα επέτρεπαν την άμεση τους χρήση χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω σχεδιασμός καθόλου για να καθησυχάσουν όσους ανησυχούσαν οι δήμαρχοι της Αμερικανικής Διάσκεψης Δημάρχων οργάνωσαν μία διάσκεψη με, όπου διέθεσαν στο ίντερνετ όλα τα έτοιμα σχέδια και έγραψαν μία έκθεση 350 σελίδων που ανέφερε 20.000 τέτοια προγράμματα από το σχεδιασμό καινούριων στολών για τους αστυνομικούς μέχρι προγράμματα δημόσιας στέγασης. Κάθε πρόγραμμα είχε το περιγραφικό του όνομα, το κονδύλιο που του είχε διατεθεί και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα δημιουργούσε. Η συνάδελφός μου Αιλίν Νόρκρος μου έδωσε την έκθεση αυτή. Την είχε ήδη μελετήσει γραμμή προς γραμμή με ένα μαρκαδόρο είχε χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος και πολλές φορές δεν μπορούσε να καταλάβει απλώς από το όνομα του προγράμματος περί τίνος ακριβώς επρόκειτο και αν άξιζε τον κόπο να χρηματοδοτηθεί. Ήξερε όμως να χρησιμοποιεί την τεχνική του crowdsourcing και με ρώτησε αν δεν μπορούσα να κάνω κάποια εφαρμογή για να το αναπτύξω. Είχε δίκιο. Άρχισα λοιπόν να δημιουργώ αυτή την εφαρμογή. Είχα ήδη εμπειρία από ιστοσελίδες, αλλά εδώ χρειαζόταν προγραμματισμός που εγώ δεν διέθετα μεταξύ των προσόντων μου. Γι' αυτό άρχισα να χρησιμοποιώ μια ήδη γνωστή τεχνολογία, το blog. Όπου είχα ζητήσει, είχα γράψει ότι ζητώ προγραμματιστές. Δύο μου απάντησαν αμέσω, δεν του γνώριζα προηγουμένω. ο Πίτερ Σνάιντερ και ο Κέβιν Ντάουιερ. Αλλά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεννοηθήκαμε και δημιουργήσαμε μαζί την ιστοσελίδα μας Stimulus Watch, τις διακοπές των Χριστουγέννων. Και στις 2 Φεβρουαρίου του 2009 λειτουργούσε. Το Stimulus Watch είναι πολύ απλό. Δηλαδή, πήραμε την έκθεση των δημάρχων και όλα τα προγράμματα τα βάλαμε στην τράπεζα δεδομένων μας. Μπορούσε λοιπόν ο πολίτης να έρθει στην ιστοσελίδα να δει το όνομα της πόλης του και να δει τι προγράμματα επρότεινε η τοπική αυτοδιοίκηση για αυτήν. Και επειδή όλα αυτά υπήρχαν στην, ε, στο ίντερνετ μπορούσε να τα μάθει ο χρήστης και ανάλογα με διάφορα κριτήρια, τίτλους, χρονολογίες κτλ και μόλις διάλεγε κάποιο χτυπούσε επάνω και του άνοιγε μία σελίδα με λεπτομερή περιγραφή. Τρία πράγματα ακόμη μπορούσε να κάνει ο χρήστης. Πρώτον, να ψηφίσει αν ενέκρινε ή όχι το πρόγραμμα. Το ερώτημα που του ετίθετο ήταν, είναι ζωτικό αυτό το πρόγραμμα και μπορούσε να απαντήσει ναι ή όχι. Ο λόγος είναι γιατί ο πρόεδρος Ομπάμα είχε υποσχέθει ότι τέτοια προγράμματα δεν θα εφαρμόζονταν παρά μόνο για ζωτικού ενδιαφέροντος θέματα, για να μην υπάρξει σπατάλη. Η ερώτηση ήταν τελείως ουδέτερη. Και η ιστοσελίδα έδειχνε αμέσως τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Δεύτερον, κάθε πρόγραμμα είχε συνοδευόταν και από μία σελίδα wiki γιατί πολλές φορές ο τίτλος μόνος του δεν ήταν πολύ περιγραφικός. Παραδείγματο χάρη, μπορεί να υπήρχε ένα πρόγραμμα μισού εκατομμυρίου δολαρίων που να λέγεται απλώς Cincinnati Street Network. Και κάποιος σαν τη συνάδελφό μου Αιλίν που δεν γνώριζε την πόλη αυτή του Cincinnati, δεν γνώριζε τι μπορεί να ήταν αυτό το πρόγραμμα. Οι πολίτες όμως της πόλης γνώριζαν ποιο ακριβώς ήταν το πρόγραμμα. Το Wiki λοιπόν επέτρεπε σε οποιονδήποτε να γράψει και να δημοσιεύσει περιγραφές και πληροφόρηση για το πρόγραμμα. Και αυτά είναι ουδέτερα πολιτικός. Είδαμε εκατοντάδες σελίδε να δημιουργούνται για τις περιγραφές αυτών των προγραμμάτων. Με τεράστιες περιγραφές. Καμία οργάνωση από μόνη της δεν θα μπορούσε να έχει χορηγήσει τόσο πολλή πληροφόρηση για τόσα πολλά προγράμματα σε τόσο λίγο χρόνο. Τρίτον, Κάθε πρόγραμμα περιείχε και μία σελίδα σχολείων όπου οι πολίτες μπορούσαν να συζητούν το πρόγραμμα. Ήταν ένα βήμα πολιτών δηλαδή, αλλά επίσης χρησιμοποιούνταν και σαν μέσο πίεσης ώστε οι πολιτικοί να μην ανακατευτούν σε τέτοιου είδους προγράμματα. Η ιστοσελίδα ήταν πολύ επιτυχής. Δύο εκατομμύρια επισκέψεις τον πρώτο μήνα. Οι σελίδες Wiki πολλαπλασιάστηκαν για πολλά προγράμματα και άρχισαν πολλές συζητήσεις. Και το πιο σημαντικό ήταν η ψηφοφορία. Μπορούσε κανείς να ελέγξει τα προγράμματα ανά αριθμό ψήφων. Μπορούσε ένας πολίτης να πει δείξτε μου τον κατάλογο των δημοφιλεστέρων προγραμμάτων. Και αυτό μπορούσε να γίνει σε επίπεδο ολόκληρης της χώρας, μίας πολιτείας ή μίας μόνο πόλης. Πάνω πάνω έβρισκε κανείς τα προγράμματα που ήταν είχαν κριθεί ως δημοφιλέστερα και από κάτω τα αντίθετα. Μετά από λίγες ώρες από τη δημιουργία της ιστοσελίδας ανάλογα προγράμματα έγιναν και για γήπεδα γκολφ, για γήπεδα άθλησης κλπ. Μερικά προγράμματα που στην αρχή φαίνονταν ανάξια χρηματοδότησης τελικά έτυχαν μεγάλης προσοχής από τους πολίτες και με τη συνάδελφο Αιλίν Νόρκρος καταλάβαμε ότι αυτό που μπορούσαν να κάνουν τα εκατομμύρια πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα μπορούσε να γίνει πολύ πιο γρήγορα από ότι από έναν ή δύο ανθρώπους. Τελικά πέρασε το νομοσχέδιο Recovery Act και θεώρησε ως απαραίτητη προϋπόθεση να είναι διαφανής η χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Εδώ ανακατεύθηκε και ο κύριος Ντεβέινι που σας μίλησε προηγουμένως. Τον Οκτώβριο του 2009 ο ιστότοπος recovery.gov άρχισε να δείχνει ποια χρηματοδοτήσεις χορηγούνταν πρώτες. Το όνομα του προγράμματος, διευθύνσεις των υπευθύνων και πολλές φορές και περιγραφές του προγράμματος. Αρχίσαμε αμέσως την δεύτερη εκδοχή του Stimulus Watch με σκοπό τον ίδιο πάλι, δηλαδή να, δώσω, να, κάνουμε, να χορηγήσουμε την ίδια εξυπηρέτηση που είχαμε κάνει με το προηγούμενο Stimulus Watch, αλλά τώρα συνοδευόμενο και από την εγκεκριμένη χρηματοδότηση και όχι μόνο τις προτάσεις, τα σχέδια προγραμμάτων. Σήμερα ο πολίτης μπορεί να τα δει όλα αυτά και η χρήση του ιστοτόπου μας είναι ανάλογη με του Recovery Gov αυτό όμως που προσθέτουμε εμείς και που δεν το δείχνει στο σελίδα Recovery.gov είναι το crowdsourcing και η συμμετοχή των πολιτών. Γιατί επαναλαμβάνω εδώ μπορούν οι πολίτες να προσθέσουν wikis για περισσότερη πληροφόρηση για κάθε πρόγραμμα. Και φυσικά μπορούν και να ψηφίζουν. Ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι ότι το crowdsourcing θα βελτιώσει την λογοδοσία και ο κύριος Ντεβέινι και οι άλλοι αυτό προσπαθούν να κάνουν. Ελπίζω η ιστοσελίδα μας να συνεισφέρει σε αυτό. Γιατί ο καθένας, ο κάθε πολίτης γνωρίζει καλύτερα αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι η λογοδοσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του crowdsourcing αλλά και ότι ανεξάρτητα προγράμματα όπως το Stimulus Watch μπορούν να βοηθήσουν. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι απλώς διαφανής η λειτουργία της κυβέρνησης, αλλά να διαθέτει και τα στοιχεία. Γιατί χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Stimulus Watch 2. Αλλά τα στοιχεία που χορηγεί πρέπει να είναι και αξιόπιστα βέβαια για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι ερευνητές. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και αναμένω τις απορίες. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα ε, η παρουσίαση και των δύο και περνούμε τώρα στη ε, συζήτηση με τους βουλευτές. Το λόγο ζήτησε ο συνάδελφος κύριος Μπάρτ Στάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω ολόψυχα τους δύο μιλητές. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπανε, γιατί δεν δουλεύει, το μικρόφωνο βεβαίω. Μια χαρά. Λοιπόν, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτά που μας είπατε. Θα πάω οπωσδήποτε και στις ιστοσελίδες να ρίξω μια ματιά ε, προς επίρρωση των όσων είπατε, γιατί πραγματικά είναι υποστηρικτικά. Έχω μερικές ερωτήσεις τώρα όμως. Πρώτον, ο νόμος του 2009, Recovery Act. Για πόσα χρήματα μιλάμε, για να καταλάβουμε έτσι, την τάξη μεγέθους και πόσα είναι τα projects, τα έργα που καλύπτονται. Γιατί σας ρωτάω, διότι εδώ συζητάμε για τα διαρθρωτικά ταμεία, το κοινωνικό ταμείο, το ταμείο συνοχής, το περιφερειακό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δεκάδες ε, χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες οι δικαιούχοι και σας ρωτώ έτσι ποια είναι η τάξη μεγέθους για να έχουμε στο μυαλό μας ε, λίγο την αναλογία. Μιλήσατε επίσης για μια ιστοσελίδα φιλική προς το χρήστη όπου όλοι οι δικαιούχοι επίσης να συμμετέχουν και πάλι πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και είναι δεδομένη η πλήρης διαφάνεια και ως προς τα δεδομένα και τι γίνεται με την ιδιωτική ε, ζωή και την προστασία στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ αυστηρή νομοθεσία για την προστασία ε, της ιδιωτικής ζωής. Ας πούμε, στο Ταμείο για τη Γεωργία, τα χρήματα που δίνονται σε αγρότες και στον κλάδο των τροφίμων ε, αναφέρονται σε μια ιστοσελίδα. Δύο Γερμανοί αγρότες διαμαρτυρήθηκαν και προσέφηγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ο εισαγγελέα δίνει μια πρώτη γνωμοδότηση και λέει ότι δεν μπορούν να δημοσιεύονται τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουμε νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Στην Αμερική τι γίνεται. Μπορείτε να δημοσιεύετε ό,τι θέλετε, τα πάντα και να είναι προσβάσιμα σε όλους. Στη συνέχεια, έχω μια ειδική ερώτηση για τον κύριο Ντέβενη. Μιλήσατε για 13 γενικού επιθεωρητές και εκείνο είναι ο πρόεδρος, αλλά υποθέτω ότι από πίσω υποστηρίζεται από μια υπηρεσία. Έχετε υπαλλήλου. Πόσοι είναι αυτοί και ποιο είναι το καθεστώ τους και πώς διασφαλίζεται στην έρευνα η ανεξαρτησία τους. Πώς συνεργάζεστε στις υπηρεσίες σας και πώς ρυθμίζεται αυτό με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, ας πούμε, τη δικαιοσύνη, την αστυνομία, το τελωνίο, την εφορία. Πώς γίνεται εκεί η διακλάδωση και η συνεργασία, γιατί είναι σημαντικές οι υπηρεσίες του κράτους και αυτές. Και τέταρτη ερώτηση. Μιλήσατε για ε, γενικούς επιθεωρητές, αλλά είναι πολίτες. Δηλαδή, πάνε και κοιτάνε την ιστοσελίδα σας και λέει εδώ κάτι πάει στραβά και το δηλώνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έτσι συχνό, δραστηριοποιούνται πολίτες ή μια φορά στο τόσο. Είναι κάτι που έχει γίνει θεσμός στη συνείδηση του κόσμου. Ε, είναι αντανακλαστικό ή θεωρητικό ότι εντάξει μπορεί και κάποιος να το καταγγείλει ε, όποτε προκύψει και αν προκύψει. Και μια τελευταία ερώτηση. Πολύ ωραία αυτά που μας είπε ο κύριος Μπρίτο, πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ενθαρρυντικά για εκείνους που θέλουν να το ψάξουν και μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο ε, για κάποιον που θέλει με κριτικό μάτι να κοιτάξει τι γίνεται με τα δημόσια κονδύλια. Αλλά θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η σχέση μεταξύ του Stimulus Watch από τη μια και της επίσημης ε, υπηρεσίας του κυρίου Ντέβανη. Έχετε καμία σχέση, συνεργάζεστε, ε, ακούει ο ένας τον άλλον, πώς γίνεται και αυτή. Ε, Ανδρέασεν. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση προς τον κύριο Ντεβάνη. Μιλήσατε για την ιστοσελίδα όπου οι δικαιούχοι αναφέρουν ε, τα χρήματα που παίρνουν και πώς αυτά μπορούν να ανακτηθούν. Μα πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι μια τέτοια ιστοσελίδα όταν οι ίδιοι δικαιούχοι αναφέρουν και όχι οι οργανισμοί πληρωμής. Κανονικά αυτοί δεν θα πρέπει. Δεν έχει άλλο τρόπο η εφορία να ψάξει ε, πώς ε, δαπανώνται τα κονδύλια και θα πρέπει να επαφιέται στον πατριωτισμό των δικαιούχων. Δεν θα πρέπει ο οργανισμός πληρωμών να τα δηλώνει αυτά ή το κράτος το ίδιο. Godmans. Ευχαριστώ. Είμαι μόνιμος εισηγητής της ε, Επιτροπής Προϋπολογισμού για τη διαχείριση των διαστατικών ταμείων. Μια ερώτηση. Στην Ευρώπη είναι διαφορετικό το σύστημα. Πληρώνουμε βασικά ε, βάση της αποζημίωσης. Βέβαια εξαρτάται από τα ταμεία, αλλά είναι επιστροφή το ποσών, αποζημίωση. Γιατί οι δικαιούχοι πληρώνουν πρώτα εκείνοι και μετά τους αποζημιώνει η κυβέρνηση και όταν έχει πληρώσει η κυβέρνηση ελέγχουμε όλα τα στοιχεία, την ε, τεκμηρίωση κτλ. Και, και δίνεται επιστροφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξ όσων γνωρίζω λοιπόν, και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τι θα κάνετε εσείς, εάν ενημερωθείτε για μία απάτη. Τι θα κάνετε, ποιον ενημερώνετε εσείς. Κάποιες αρχές, κάποιον οργανισμό για την αποτελεσματική... Όχι, δεν μιλώ για την απάτη, συγγνώμη, διορθώνει ο μιλήτης όταν είναι χαμηλή απορρόφηση, όταν δεν καλύπτουν τα πλάνα τους, όταν δεν απορροφούν τα κονδύλια και δεν ε, ενεργούν σωστά οι δικαιούχοι. Τι κάνετε, ποιον ενημερώνετε, αν ενημερώνετε κάποιον. Δεν μιλάω για απάτη. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτό που ακούσαμε. Έχω μερικές ερωτήσεις στον κύριο Ντεβάνη. Είπατε ότι βάλετε λάθος στοιχεία. Αν, βάλετε, ε, ε, αν, σας δίνουν λάθος στοιχεία, τι γίνεται. Ζητάτε αποζημίωση, πόσο κοστίζει το σύστημα αυτό και ποιε είναι οι διοικητικέ δαπάνες και ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται. Είπατε ότι κάθε τρίμηνο δικαιούχο αναφέρει ηλεκτρονικά. Με ποια πειθαρχία και πώς τον υποχρεώνεται, ποια είναι τα πρόστιμα και ποιε είναι οι απαιτήσει για την ανάκτηση και ποια είναι η διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση ή απλώς μια διοικητική απόφαση ε, που μπορεί ε, να αξιώνει ε, την επιστροφή χρημάτων. Και πώς γίνεται ο έλεγχος και πώς μετράτε την επιτυχία του ελέγχου. Για σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα σε διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης, όταν ε, ε, οι δικαιούχοι δημοσιεύονται, τους εκβιάζουν και τους πουλάνε προστασία ορισμένα εγκληματικά δίκτυα. Στην Αμερική συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις για έργα δημόσια, ε, τα οποία ο κόσμος αφισβητεί στο διαδίκτυο. Ας πούμε, εγώ αγωνίζομαι για διάφορα έργα και λογοδοτώ, αλλά δεν θέλω να είμαι υποπίεση. Και εγώ ε, το βλέπω αυτό και ως μια πίεση. Τι κάνουν ε, οι βουλευτές της Ηνωμένε Πολιτείε ε, σε αυτή την περίπτωση όταν τους πιέζουν. Ευχαριστώ. Βάουγκρ. Yeah, uh, Um, the... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαδικασία που μας περιγράψατε σήμερα το πρωί είναι πολύ εντυπωσιακή. Δεν ξέρω αν κάποιε από τι περιφέρειες που ασχολούνται με τα που λαμβάνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν ένα τόσο εκτεταμένο σύστημα να το εφαρμόσουν. Λόγω χάρη στην Ουαλία έχουμε ένα εξαιρετικό ιστότοπο, ο οποίο καλύπτει όλα τα προγράμματα για τα οποία υποβάλλονται αιτήσει και για τα οποία λαμβάνουμε χρηματοδότηση. Αλλά δεν φτάνει το εύρο του δικού σα ιστοτόπου. Τώρα, για την κλίμακα των ζητημάτων που σας απασχολούν στις ΗΠΑ. Εμείς, μάλλον εσείς έχετε μπορέσει να δείτε το ποσοστό των προγραμμάτων ε, για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσει και που μπορεί να έχουν σχέση με απάτη και καταπολέμηση και κακοδιαχείριση, εσείς κάνατε διάκριση μεταξύ ε, απάτης και σφαλμάτων στο σύστημά σας. Και επίσης για τον υψηλό κίνδυνο. Είναι μηδενική η ανοχή σας ως προς την απάτη ή δέχεστε ένα τάδε ποσοστό προγραμμάτων που μπορεί να έχουν και ένα μέρος κινδύνου, λόγω χάρη. Και επίσης για τις κατηγορίες που μπορεί να διατυπώνονται στα διάφορα στους ιστοτόπους και τους δύο που παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί. Είδαμε ότι κάποιε φορές υπάρχουν ομάδε συμφερόντων, εκπροσώπων συμφερόντων ή μεμονωμένε κατηγορίες που μπορεί να απευθύνονται για συγκεκριμένου λόγους για να ασκηθούν πιέσει. Εσεί, Εσείς λοιπόν πώς ε, ασχολείστε με τις ψευδεί κατηγορίες, πώς τις κάλυπτετε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σόνεγκάρτ. Øh, øh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε για, για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που ακούσαμε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν ε, εντοπίζονται ατασταλίες ή ε, περίπτωσης απάτης, ποιες είναι οι διαδικασίες ανάκτησης που εφαρμόζονται. Επίσης, έχετε στατιστικά στοιχεία κύριε Ντβέινη. Και αυτό έχει σχέση και με το προηγούμενο ερώτημα. Στατιστικά στοιχεία για την αναλογία πιστώσεων που εκταμιεύονται και κακώς δαπανούνται, κακοδαπανήθηκαν λόγω απάτης ή λόγω σφάλματος ή παραβλεψίας. Ε, υπάρχει διαφορά μεταξύ σφάλματος και απάτης. Τι στατιστικά στοιχεία υπάρχουν λοιπόν να καθορίσετε ποσοστά. Και επειδή είσαστε επικεφαλής αυτού του συμβουλίου, φαντάζομαι ότι κάτι θα έχετε να μας πείτε για αυτό το θέμα. Ο κύριος Δεμπρίτο τώρα. Κατανοώ ότι μπορεί κανείς με τον ταχυδρομικό του κώδικα να έχει πρόσβαση στο σύστημα, πληκτρογόντας απλώς αυτόν τον κωδικό. Όμως μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μόνο τα τοπικά προγράμματα ή το σύνολο των προγραμμάτων που περιλαμβάνει ο τόπος και έχουν κλίμακα εθνική. Ευχαριστούμε ο Γκάγερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ και τους δύο κυρίους για τα όσα μας είπαν. Έχω μια ερώτηση και με κάλυψε ο συνάδελφος Σόναγκαρτ. Δεν θα την κάνω. Αλλά έχω άλλη ερώτηση στον κύριο Ντέβανη. Μήπως δεν το κατάλαβα σωστά. Είπατε ότι οι περιφέρειες των Ηνωμένων Πολιτειών όπου η κρίση ε, σώβησε ιδιαίτερα θεωρείται παράγον κινδύνου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί το ταξινομείται αυτό ως παράγοντα κινδύνου, επειδή κάποιες περιοχές επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Και άλλη μια ερώτηση για την ένταση που υπάρχει ανάμεσα στα ιδιωτικά στοιχεία και τη δημόσια πληροφόρηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κάναμε τέτοιες προτάσεις, θα ήμουν βέβαιος εγώ ότι διάφορες οργανώσεις συμφερόντων ε, επιχειρήσεων ε, θα απέρριπταν αυτά γιατί θα σου λέγει υπάρχει το εμπορικό απόρριτο, είναι στοιχεία εμπιστευτικά για την κατάσταση της ρευτότητας της επιχείρησης, για την καινοτομία, για κάποια σχέδια είναι βιομηχανικά απόρριτα, αυτά εμπορικά απόρριτα και θα το απέριπταν. Και ως βουλευτές θα είχαμε πρόβλημα να ε, τακμηριώσουμε αυτά τα επιχειρήματα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στι Ηνωμένε Πολιτείε πώς το έχετε λύσει αυτό το θέμα για τους δικαιούχους, στο βαθμό που είναι επιχειρήσεις. Σου λέει δεν μπορώ να αποκαλύψω τα μυστικά της επιχείρησης. Ε, πολύ ωραία υποχρέωση για ενημέρωση, αλλά πού σταματάει η ενημέρωση. Grazie. Ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τώρα τους ε, μιλητές μας, τον κύριο Ντέβιν πρώτα. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το σύνολο του ποσού, τα 787 δις δολάρια. Έως τώρα, περίπου 175.000 δικαιούχοι έχουν ε, εντοπιστεί για τα κονδύλια αυτά. Τα έχουμε, τους έχουμε διαιρέσει σε δύο κατηγορίες, τους βασικούς δικαιούχους που πρώτοι θα πάρουν τα κονδύλια και τους δευτερο, δευτερεύοντες. Τους ονομάζουμε subprimes, εκείνοι που θα πάρουν σε δεύτερη φάση χρηματοδότηση. Όλοι αυτοί οδηγούν σε αυτό το τελικό αριθμό. Περίπου 29 υπηρεσίες κυβερνητικές υπάρχουν στις ΗΠΑ που συγκεντρώνουν αυτά τα κονδύλια για να τα μοιράσουν στους δικαιούχους. 29 λοιπόν γενικοί επιθεωρητές, οι οποίοι είναι έτοιμοι, αν τους το ζητήσουμε, να προχωρήσουν σε έρευνες και έλεγχο για τα κονδύλια. Οπότε και εμείς ενισχύουμε τους πόρους μας μέσω της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και έχουμε το δικαίωμα ως Συμβούλιο να ζητήσουμε από τους γενικούς επιθεωρητές να κάνουν τέτοιου είδους έρευνες και έλεγχους. Και οι αρχές μπορούν να το κάνουν και με δική τους πρωτοβουλία. Λόγου χάρη, ως τώρα, έχουμε κάνει τουλάχιστον 500 ελέγχους και περίπου 300, 450 ποινικέ έρευνες έχουν διεξαχθεί. Έχουν ξεκινήσει μάλλον σε όλη τη χώρα. Οπότε έχουμε ένα μικρό αριθμό στο προσωπικό του Συμβουλίου στη Washington, 50 άτομα περίπου. Και ενισχύουμε και τους υπόλοιπους 29 γενικούς επιθεωρητές. Ίσως να είναι και 8.000 οι εργαζόμενοι σύνολο, ερευνητέ και γενικοί επιθεωρητέ μαζί. Έχουμε λοιπόν το απαραίτητο προσωπικό για να φέρουμε το καθήκον αυτό. Τώρα, ε, μιλήσατε και για τους πολίτες γενικούς επιθεωρητές, όπως τους ονομάζουμε κάποιοι. Θα περίμεναν ότι θα υπήρχαν εκατομμύρια τέτοιοι πολίτες, αλλά αυτό ήταν ίσως κάπως περισσαόδοξο ως πρόβλεψη. Σε κάθε περίπτωση, εκατοντάδες πολίτες μας ε, ειδοποιούν κάθε μήνα και έχουμε ένα πολύπλοκο σύστημα ελέγχου αυτών των ε, τηλεφωνημάτων ώστε να απομακρύνουμε τα τηλεφωνήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα θέματά μα. Κάποιοι τηλεφωνούν για να παραπονηθούν για τον πρόεδρο Ομπάμα, την κυβέρνηση, οτιδήποτε του περνάει από το μυαλό και κοιτάζουμε να κρατήσουμε τα τηλεφωνήματα, τι επαφέ που έχουν ε, μεγαλύτερη σχέση με την απάτη και τη σπατάλη. Είναι περίπου ένα στα δέκα. Αυτή ήταν η πείρα μου τις τελευταίες δεκαετίες και στη, στο επίπεδο των πυρεών καταστολής. Δίωξη μάλλον. Ε, ένα στα δέκα τηλεφωνήματα έχουν σχέση με κάποια σοβαρή υπόθεση έρευνα. Οι υπόλοιποι είναι απλώ θυμωμένοι, παραπονιούνται ή θέλουν να μιλήσουν σε κάποιον γιατί έχουν κάποιο προσωπικό πρόβλημα στη μέση τη νύχτα. Έχουμε πάντω ένα πολύπλοκο σύστημα με τηλεφωνητέ, με ερωτηματολόγια, αυτό μπορεί να γίνει και με τηλέφωνο, με φάξ ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Μπορεί κανεί να υποβάλει τι παρατηρήσει του για περιπτώσεις πατάλης ή απάτης. Τώρα, πώς ε, λαμβάνουμε δεδομένα για τους δικαιούχους και πώς διαχωρίζουμε τους δικαιούχους από τους φορείς. Σε κάθε περίπτωση συγκεντρώνουμε και τα δύο. Πρώτα απ' όλα συλλέγουμε δεδομένα για δικαιούχους, δηλαδή για αυτούς που έχουν πάρει κονδύλια και για να απαντήσω και ένα ερώτημα που τέθηκε αργότερα, όλοι οι δικαιούχοι των κονδυλίων της ανάκτησης που εμείς παρακολουθούμε, είναι φορείς, είναι ενώσεις, δεν είναι άτομα. Οπότε εδώ δεν μιλούμε για ζητήματα ιδιωτικού βίου σε σχέση με τα δημόσια κονδύλια, που μπορεί να μιλάμε για κονδύλια που απευθύνονται σε επιχειρήσει, σε ενώσει. Οπότε παίρνουμε πληροφορίε από εταιρείε για το τι έκαναν τα κονδύλια. Και σε κάθε περίπτωση δεν παραβιάζουμε του νόμου ιδιωτικού βίου των ΗΠΑ. Ιδάλλως θα είχε πάση τη λειτουργία του το Συμβουλίο μας, πολύ νωρίτερα. Παρακολουθούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτά τα δημόσια κονδύλια και θεωρούμε ότι σε σχέση με δημόσια κονδύλια δεν μπορεί να τίθενται ζητήματα ιδιωτικού βίου. Εάν λαμβάναμε στοιχεία για ιδιώτε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Για τι πληροφορίε τώρα σε σχέση με του οργανισμού. Κοιτάζουμε σε ποιον έδωσαν τα κονδύλια. Φαντάζομαι ότι δεν θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιες φορές έχουμε προβλήματα μέχρι να καταλάβουμε και να εντοπίσουμε σε ποιον έδωσαν τα χρήματα οι οργανισμοί και οι φορείς. Και εκείνοι δυσκολεύονται να μας δώσουν στοιχεία. Όσο και οι δικαιούχοι για το τι έκαναν με τα χρήματα. Εμείς πρέπει να κάτσουμε και να διασταυρώσουμε τα στοιχεία. Τις πληροφορίες που έρχονται από τους οργανισμούς και τους φορείς και αυτά που μας λένε οι πολίτες δεν είναι πάντοτε απόλυτη αντιστοίχηση, αλλά καταφέρνουμε να βελτιωθούμε με τους κύκλους υποβολής εκθέσεων και οι δικαιούχοι αρχίζουν να συνηθίζουν την καταγραφή των στοιχείων. Από τις πληροφορίες που ζητούμε βάσει αυτού του συστήματος υπάρχουν τουλάχιστον 99 διαφορετικά ε, στοιχεία που ζητούνται οι πολίτες να συμπληρώσουν, καθώς και οργανισμοί, ώστε να μας πούν τι έγινε με τα κονδύλια. Τώρα, όταν εντοπίζουμε περιπτώσεις απάτησης πατάλη, ε, το αναφέρουμε στον Γενικό Επιθεωρητή της υπηρεσία που έδωσε τα κονδύλια. Δηλαδή, ένα σχέδιο κατασκευής δρόμου, με πληροφορίες από πολίτες ή ερευνητών που εντόπισαν κακοδιαχείριση. Αμέσως το θέμα παραπέμπεται στην, στο Υπουργείο Μεταφορών ή την Υπηρεσία Μεταφορών και γενικό Διευθυντής φροντίζει τον έλεγχο ή την έρευνα και φροντίζει να ενημερώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Και εκείνοι αποφασίζουν εάν θα γίνει δίωξη ή όχι. Εάν υπάρξει δίωξη, κάποιε φορέ τα χρήματα επιστρέφονται. Άλλοτε υπάρχει αστική διαδικασία για να επιστραφούν τα χρήματα. Πάντως, στην ομιλία μου περιέγραψα τρόπους να προλάβουμε το να συμβεί απάτη, να έχουμε υπόθεση απάτη σε κάθε περίπτωση. Το να έρθει κανεί μια διετία αργότερα για να διαπιστώσει ότι λείπουν χρήματα δεν είναι επιτυχία. Η επιτυχία μα μετράται από την πρόληψη τη απάτη. Και διαρκώ ως προς τη χρήση των τεχνολογιών και των τεχνικών που ανέφερα προηγουμένως, ε, εξευρίσκουμε περιπτώσεις απάτης ή σπατάλης εγκαίρως. Οπότε καλούμε αμέσως το φορέα την υπηρεσία που δίνει τα κονδύλια και λέμε σταματήστε να χρηματοδοτείτε αυτόν τον δικαιούχο. Δείτε πώς δαπανώνται και μετά ε, συνεχίστε, ζητήστε τα πίσω. Και έτσι γίνεται έλεγχος. Η, σπαταλης οποτε καλουμε αμεσως το φορεα την υπηρεσια που δινει τα κονδυλια δίωξη αναλόγως στην περίπτωση. Όπως αναφέρθηκε, έχουμε αρκετά σφάλματα στα δεδομένα μας την πρώτη φορά που αρχίσαμε να συλλέγουμε δεδομένα ιδίω, προφανώς ζητούσαμε από τους υπευθύνου των εταιριών να μας ενημερώσουν για πρώτη φορά για περισσότερα δεδομένα από όσα ποτέ του είχαν ζητηθεί. Υπήρχαν λοιπόν πολλά ασφάλματα στα δεδομένα. Τη δεύτερη φορά, στο δεύτερο κύκλο υποβολή εκθέσεων, υπήρχαν σαφώ λιγότερα ασφάλματα. Και τώρα, στον τέταρτο κύκλο, με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να σα πω ότι έχουμε ακόμη λιγότερα ασφάλματα από ό,τι ποτέ στο παρελθόν. Και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε κι άλλο όσο περνάει ο καιρό. Και όσο συνηθίζουν και οι υπεύθυνοι στην ε, συλλογή των στοιχείων. Το σύστημα υποβολή εκθέσεων που περιέγραψα νωρίτερα είναι ένα ξεχωριστό ιστότοπο. Ε, προστατεύεται με κωδικό πρόσβαση. Και εκεί μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε αυτά που ονομάζουμε logic models, ε, λογικά πρότυπα και με σύστημα ελέγχου για να αποτρέπουμε τα σφάλματα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στην πρώτη περίοδο υποβολή εκθέσεων ε, δεν έβαζαν το σωστό τμήμα περιοχής, το σωστό κωδικό περιοχής για να φανεί ποιον εκπροσωπούν αυτοί που συμπληρώνουν τα δεδομένα. Αυτό θύμωνε τα μέλη του Κογκρέσου. Έβλεπαν να μην καταγράφονται σωστά οι περιοχές. Οπότε υπήρχαν σφάλματα. Έτσι λοιπόν έβαζαν ένα τυχαίο αριθμό στο σύστημα οι... αυτοί που συμπληρώναν τα στοιχεία για... και δεν μπορούσαν να περάσουν σωστά στις επόμενες ερωτήσεις. Τώρα προλαμβάνουμε το σφάλμα αυτό με τον ταχυδρομικό κώδικα. Εάν ο ταχυδρομικός κώδικας δεν συνδυάζεται με τον κωδικό της περιοχής, πρέπει να, μείνει, να διαλέξουν αυτοί που συμπληρώνουν τα στοιχεία. Τέλος πάντων αυτό το έχουμε επιλύσει υποδεικνύοντας το σωστό αριθμό στην οθόνη. Προσαρμόζουμε δηλαδή και εμείς το σύστημα στο να μπορούμε να περιορίζουμε το να συμβαίνουν τέτοια σφάλματα. Τώρα, κυρώσει ή για μη υποβολή στοιχείων. Δυστυχώ, όταν το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο για την ανάκτηση, δεν προέβλεψε κυρώσει για τη μη υποβολή στοιχείων. Στον πρώτο κύκλο υποβολή στοιχείων βρήκαμε περίπου 4.000 δικαιούχου που δεν είχαν υποβάλει στοιχεία. Ο αριθμό αυτό έχει μειωθεί τώρα σε περίπου χίλιους. Και εκείνοι που δεν υπέβαλαν στοιχεία τρει ή περισσότερε φορές είναι μόνον 31. είναι εκείνοι που, για τους οποίους δεν έχουμε καθόλου στοιχεία και βεβαίως εκεί θέλουμε να πάυσουμε τη χρηματοδότηση και να πάρουμε πίσω τα κονδύλια, εφόσον δεν δαπανήθηκαν. Πολλά χρήματα επίσης έχουν αποδοθεί χωρίς να έχουν ε, δαπανηθεί, οπότε μπορούμε να τα πάρουμε πίσω. Δεν έχουμε επίσης δει ενδείξεις αργων, δράσεων οργανωμένου εγκλήματος, εγκληματικών οργανώσεων σε σχέση με αυτά τα κονδύλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει, απλώς δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Θα είχαμε όμω δει κάποιο δείγμα, φαντάζομαι, τέτοιων τάσεων. Και σίγουρα θα υπάρχουν και περιπτώσεις διαφθοράς, καθώς οι τοπικοί θύνοντες κάπως έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια, είναι αναπόφευκτο κάτι τέτοιο, ξέρουμε ότι θα συμβεί Έχουμε κάποιε ποινικέ υποθέσει που εκδικάζονται αυτή τη στιγμή και έχουν σχέση με δημόσια διαφθορά. Όμω υπάρχει πολλή πίεση προ όλου, ώστε να διαβεβαιωνόμαστε ότι δεν θα συμβαίνουν τέτοια τι περιπτώσει. Η διαφάνεια σε αυτή την περίπτωση έχει στρέψει το βλέμμα όλων σε αυτά τα, σε κονδύλια. Οι, οι ε, αποφεύγουν αυτά τα κονδύλια, όσο στρέφονται αλλού. Εγώ αν ήθελα να κλέψω, δεν θα πήγαινα να κλέψω από αυτά τα λεφτά. Όλοι παρακολουθούν τι γίνεται με αυτά τα κονδύλια. Οι πολίτε, οι δημοσιογράφοι καθημερινά πηγαίνουν στον ιστότοπο και προσπαθούν να εντοπίσουν προβλήματα. Ε, εάν έχουν πάει τα κονδύλια σε ανθρώπου που δεν έπρεπε να τα λάβουν. Οι πολιτικοί σε, όλη, τη χώρα, οι ομοσπονδιακοί, οι τοπικοί, οι δήμαρχοι, οι τοπικοί άρχοντε, όλοι παρακολουθούν πού πηγαίνουν τα χρήματα. Να είναι βέβαιοι ότι δεν έχουν κλαπεί, δεν έχουν ε, χρησιμοποιηθεί για απάτες. Είναι τα πάντα ορατά, διαφανή. Υπάρχει λοιπόν σοβαρή άσκηση πίεση και από τους πολίτες, γιατί μπορούν να κοιτάξουν από, για πρώτη φορά πώς ακριβώς δαπανήθηκαν τα κονδύλια στις ΗΠΑ. Όπως είπε και ο κύριο Μπρίτο, Εάν ε, κανείς το παρακολουθήσει προσεκτικά μπορεί να δει πως ε, έχουν ταπανηθεί τα κονδύλια. Όμως οι πολίτες θέλουν να μπορούν να βγουν και στο δρόμο τους, να δουν κατά πόσον τα προγράμματα εκτελούνται. Μια γέφυρα, ένα σχολείο, ένας δρόμος. Εάν κάτι έχει πάει στραβά, εάν δουν ότι κάποιος έχει ιδιαίτερη σχέση με ένα τοπικό άρχοντα λόγου χάρη, θα μας ε, ειδοποιήσει. Είναι λοιπόν τεράστιο το όφελο. Εγώ ε, έχω εργαστεί στη δίωξη ε, εδώ 40 χρόνια περίπου. Δεν είναι ανοιχτή αυτή η υπηρεσία. Για μένα λοιπόν ήταν μεγάλη αλλαγή να συμμετάσχω σε αυτή την μετατόπιση. Και η διαφάνεια βοηθά τη λογοδοσία, βοηθά την ε, επιβολή του νόμου. Είναι η πρώτη φορά που τόσα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτό το θέμα και ενισχύεται και η δίωξη του οικονομικού εγκλήματο τουλάχιστον σε επίπεδο ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Έχουμε μηδενική άνοχη για την απάτη. Αυτό ανακοινώθηκε και από τον Γενικό Εισαγγελέα των ΗΠΑ. Και αυτό σημαίνει ότι θα διώκεται οποιοδήποτε είναι υπεύθυνο για απάτη οπουδήποτε και για οποιοδήποτε ποσό και αν πρόκειται. Τώρα για τους παράγοντες κινδύνου που ανέφερα προηγουμένως, ίσως κάποιες εξηγήσεις. Εξετάζουμε το ιστορικό που είχαμε περιπτώσεις απάτη στο παρελθόν σε σχέση με ποια προγράμματα. Κοιτάζουμε προηγούμενες εκθέσεις που έχουν υποβληθεί από γενικούς επιθεωρητές και άλλους στο σύνολο της κοινότητας των επιθεωρητών. Βλέπουμε πού έχει πλήξει περισσότερο περιοχές η οικονομική ύφεση που ευθύνεται για κλείσιμο επιχειρήσεων και εταιριών. Κοιτάζουμε πού πήγαν τα κονδύλια, τα διασταυρώνουμε και φροντίζουμε να δούμε τις διάφορες διαστρωματώσεις. Μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε με κάποιο ποσοστό βεβαιότητας που πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν περισσότερες τάσεις για απάτη, για άλλες περιπτώσεις. Έτσι μπορούμε λοιπόν να κατευθύνουμε τους ερευνητές, τους επιθεωρητές σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές όταν μπορεί να προκύψει κάποια απάτη. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ αν έχετε και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ να παρέμβω και πάλι. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπρίτο για τις υπόλοιπες απαντήσεις. Um, so Καταρχήν, ο κύριος Ντεβέινι κάλυψε πολλά από αυτά που ήθελα να πω και εγώ. η σχέση μεταξύ του Stimulus Watch και της οργάνωσης του υπάρχει. Έχουμε εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου για μαρτυρία και να με διορθώσει ο κύριος Δεβένη αν κάνω λάθος. Η δική του δουλειά είναι κυρίως η επιβολή του νόμου. Όταν όμως εγώ δίνω συστάσεις ως προς τη βελτίωση των πραγμάτων. Τις συστάσεις αυτές τις κάνω ή στο σύνολο του Κογκρέσου ή στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και εκείνοι τις ερμηνεύουν μετά. Σε αυτό το βαθμό λοιπόν μπορώ να πω ότι έχουν ανταποκριθεί και ιδιαίτερα αυτή η κυβέρνηση επιμένει ιδιαίτερα στη διαφάνεια και ακούει περισσότερο τέτοιου είδους συστάσεις. Δεν τις εφαρμόζει βέβαια πάντοτε γιατί είναι δύσκολο να αλλάξει κανείς υπάρχοντα νομοσχέδια. Οι αναφορές όμως που κάνουν οι όσοι παίρνουν τα κονδύλια δεν είναι πάντοτε πλήρης. Υπάρχουν οι πρώτοι αποδέκτες και οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να υποχορηγήσουν κονδύλια σε τρίτον. Θα ήθελα και αυτό το επίπεδο δαπάνησης βέβαια να είναι διαφανές, αλλά δεν υπάρχει ακόμα. Και θα έπρεπε να προβλεφθούν και κυρώσεις για την μη αναφορά των στοιχείων. Κάποιες κυρώσεις τέλος πάντων κάνα προς τη μούλη. Άλλο ερώτημα που τέθηκε ήταν πώς αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι μπορεί κανείς να προσθέσει στοιχεία στην ιστοσελίδα μας. Πρώτον, αφού είναι wiki, γι' αυτό ακριβώς μπορεί ο καθένας να προσθέσει. Άρα το πρόγραμμα αυτό από μόνο του διορθώνει την δυναμική της ιστοσελίδας. Σκεφτείτε την Wikipedia. Εκεί μπορεί κανείς να προσθέσει άρθρα, να διορθώσει πληροφορίες και είναι πολύ πιο εύκολο να επανέλθει κανείς στην προηγούμενη εκδοχή παρά να διορθώσει. Άρα μπορεί κάποιος να διορθώσει επίσης κάτι που προστέθηκε λάθος, κακός. Στην πρώτη ιστοσελίδα του Stimulus Watch ζητήσαμε από τοπικές αρχές να μας πούν πώς λειτουργεί η σελίδα, μας είπαν αυτό είναι λάθος, εκείνο δεν πάει καλά και είχαμε βασιστεί ήδη από την αρχή στα λόγια της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκείνη την έκθεση των δημάρχων. Καμιά φορά μας ζήτησαν αλλαγές, αφού εξήγησαν καλά και γιατί, και τις κάναμε. Τέλος, όπως και η Wikipedia, Έχω διδάξει και εγώ φοιτητέ νομικής και δεν θα δεχόμουν ποτέ ένα φοιτητή που θα μου έλεγε τις πληροφορίες μου τις πήρα από τη Wikipedia. Δεν είναι αποδεκτή ακαδημαϊκή πηγή, αλλά ταυτόχρονα τους ενθαρρύνω να χρησιμοποιήσουν την Wikipedia γιατί είναι πολύ καλή αρχή. Δεν είναι όμως και η τελευταία λέξη όπως και για τη δική μας σελίδα, αν έχει καταψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ανάξιο λόγου. Είναι απλώς ένα θέμα έρευνας και πληροφόρησης. Τα βλέπω λοιπόν αυτά ως απλώς μια αρχή, μια βάση. Τέλος, με ρώτησαν η διαφάνεια υπάρχει σε τοπικό, όχι μόνο εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτιών. Φαίνεται ότι και σε αυτό το επίπεδο των πολιτιών γίνεται όλο και σημαντικότερη η διαφάνεια και πολλοί πολιτιακοί νομοθέτε αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες για μεγαλύτερη και περισσότερη διαφάνεια. Ακόμη και στο τοπικό επίπεδο φαίνονται αυτά για την παραδείγματο χάρη. Ακόμη και μερικά σχολεία έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν τις δαπάνες των. Υπάρχει μεγάλη πρόοδος λοιπόν, μεγάλη. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο Αμερικανούς μας ομιλητές για την πολύτιμη συνεισφορά τους στις εργασίες της Επιτροπής μας και τώρα περνάμε στην ευρωπαϊκή διάσταση της ακροασής μας. Χαιρετίζουμε την κυρία Ζουλή Πελεγκρίν που εργάζεται στο Κέντρο Βιομηχανικών Σπουδών στο Μιλάνο, είναι πολιτική επιστήμονα και θα μας μιλήσει για τα πορίσματα έρευνας που έγινε για λογαριασμό του Ευρωκοινοβουλίου με τίτλο «Η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των δεδομένων και ο αντίκτυπός της στην πολιτική συνοχής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζουλή Περεγκλέ, ναι, εκπροσωπώ το Κέντρο Βιομηχανικών ε, Μελετών του Μιλάνου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, ευκαιρία που έχω να σας παρουσιάσω σήμερα εδώ τα αποτελέσματα της μελέτης που έγινε πριν από ένα περίπου έτους για τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Διαφάνειας στην πολιτική συνοχής. Καταρχάς, σύντομα θα σκιαγραφίσω το στόχο της ε, πρωτοβουλίας αυτής για τη διαφάνεια και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια θα περάσω μια επισκόπηση τα κύρια ευρήματα της μελέτης για την οποία εφαρμόσαμε στην πολιτική συνοχή στα κράτη-μέλη και θα καταλήξω με μια μικρή σειρά συστάσεων που προέκυψαν από τις μελέτες αυτές. Λοιπόν, τον Νοέμβριο του 2005 ε, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία Διαφάνειας μετά από μια ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάλλας που ήταν αρμόδιος για θέματα διοικητικά και καταπολέμησης απάτης και ζητούσε να επανέλθει η εμπιστοσύνη και η πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε προηγηθεί το διπλό όχι στη Γαλλία και την Ολλανδία στα δημοψηφίσματα σχετικά με ε, τη συνθήκη. Ε, έλεγε λοιπόν ο Επίτροπος τότε και τα επίσημα έγγραφα ότι Στόχος είναι η νομιμότητα, η εμπιστοσύνη, η λογοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μάιο στη συνέχεια του 2006 ε, εγκρίθηκε μια πράσινη βίβλος με τέσσερα ε, βασικά στοιχεία πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, κανόνες και πρότυπα δεοντολογίας για δημοσίους υπαλλήλους, διαφάνεια των λόμπι των ομάδων συμφερόντων και ελάχιστα πρότυπα για τη διαβούλευση και διαφάνεια στη χρήση των κοινοτικών πόρων με δημοσιοποίηση των ε, δικαιούχων. Εκεί λοιπόν εστιάστηκε η μελέτη και εκεί θα εστιαστεί και η δική μου παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα διορθωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, όπως θα γνωρίζετε, είναι στη συνυπευθυνότητα. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται αυτά τα ταμεία και όχι τα κράτη-μέλη. Και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη. Τα κράτη-μέλη λοιπόν. Άρα, θα πρέπει να δημοσιεύονται τα στοιχεία αυτά. Θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιεύουμε τα στοιχεία για τους δικαιούχους. Αυτό ρωτούσαμε λοιπόν στη διαβούλευση ε, και ε, το ρωτούσε και η πράσινη βίβλος και η απάντηση ήταν ναι, ένα μαζικό ναι, αλλά με επιπλέον ε, όρους ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό. Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και ε, θέσπιση κοινών προτύπων και κανόνων για να επιτρέπεται, ε, διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το νομικό πλαίσιο, να θεωρήθηκε ο δημοσιονομικός κανονισμός και ζητούσε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη να δημοσιεύουν στοιχεία για τους δικαιούχους, για ε, το κομμάτι του προϋπολογισμού που τους αναλογούσε και ιδιαίτερα στην πολιτική συνοχής ε, υπήρχε και ξεχωριστό άρθρο στον εφαρμοστικό κανονισμό των ταμείων που όριζε και παραθέτω ότι η διαχειριστική αρχή θα είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση ε, τουλάχιστον τη εξή ενημέρωσης και των μέτρων. Δημοσίευση ηλεκτρονικά ή άλλο ε, του καταλόγου εγγυούχων, δικαιούχων, τα ονόματα των δράσεων και τα ποσά που διατίθενται στις δράσεις αυτές. Um, Σε ό,τι αφορά το κοινά πρότυπα, υπήρξε και ένα συνοδευτικό σημείωμα ε, της ε, Αρμόδιας Επιτροπής, ένα προσανατολιστικό έτσι, βοήθημα της COCOF ε, όπως ονομάζεται Αρμόδια Επιτροπή, που εντόπιζε και καθόριζε τους τομείς για συλλογή στοιχείων. Και ποια είναι αυτά, είπαμε, το όνομα, ε, του δικαιούχου το έτος, το όνομα της δράσης, ε, το έτος της τελικής πληρωμής, τα ποσά που έχουν ε, δεσμευτεί, καθώς επίσης και το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί στο τέλος της δράσης. Για ποιο λόγο. Ζητούσαμε και να δούμε ποια είναι η δέσμευση των πληρωμών για να μπουν τα στοιχεία αυτά στο πρόγραμμα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε δηλαδή την ολοκλήρωση του έργου. Τώρα, Πώς εφαρμόστηκαν όλα αυτά στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες. Δύο είναι οι πηγές των στοιχείων μας. Ε, τα στοιχεία στο διαδίκτυο έτσι πατώντας ένα κουμπί στα γραφεία μας, αλλά και, ε, και οι κατά περίπτωση ε, μελέτες σε ξεχωριστές χώρες, Φιλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Πολωνία που έχουν διαφορετική παράδοση και στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων με διάφορα ταμεία. Πρόσβαση, κατανόηση, αξιοπιστία, χρησιμότητα <laughs> και διάφορους ε, παράγοντες επεξηγηματικούς που θα αναλύσω στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόσβαση. Ζητώ συγγνώμη για τη διαφάνεια. Είναι πολύ μικρογραμμένα, αλλά έχετε στους φακέλους σας ε, τις διαφάνειες, στο έγγραφο που σας διανεμήθηκε. Αυτή είναι η σελίδα λοιπόν που βλέπετε για τη διαφάνεια που ανοίγει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν πληκτρολογήσετε διαφάνεια. Στη συνέχεια σας στέλνει στο σύστημα ε, οικονομικής διαφάνειας που αφορά ε, κονδύλια και πόρους που διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι περίπου το 20% του κοινοτικού προπολογισμού ή στη συγχρηματοδότηση και στην υπευθυνότητα ε, που διαχειρίζονται από κοινού τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχής, από τη μια Έχουμε το Ταμείο Συνοχής, το οποίο διαχειρίζεται ε, η Γενική Διεύθυνση για τις Περιφέρειες και ε, άλλα ταμεία διαρθωτικά, γεωργικό ας πούμε, που διαχειρίζεται η ε, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Αυτό μπορείτε να το ζητήσετε λοιπόν, ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ας πούμε, σας παραπέμπει μετά στα, στις περιφερειακές του σελίδες των διαφόρων περιφερειών και των δικαιούχων. Πόσα κλικ λοιπόν χρειάζονται για να φτάσουμε στα στοιχεία. Κατά μέσο όρο 1,5 για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Ταμείου και 1,9 για ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής, που εκ πρώτης όψεως δεν είναι και άσχημο αλλά δεν είναι πάρα πολύ απλό για εκείνους που δεν έχουν έτσι, μεγάλη εξοικείωση ε, της ιστοσελίδας ε, και του διαδικτύου ως προς την πολιτική συνοχή. Έτσι έχουν τα στοιχεία λοιπόν το Μάρτιο του 2009 όπως βλέπετε τώρα. Δεν είναι απολύτως ικανοποιητικά, καταλαβαίνετε. Υπάρχουν χώρες, ολόκληρες η περιφέρειες που δεν έχουν δώσει στοιχεία η Ελλάδα, η Ισπανία, μερικές περιφέρειες της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και η Αυστρία για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Βεβαίω έχουν αλλάξει τα πράγματα έκτοτε, αλλά παραμένει η κατάσταση έτσι κάπως ε, ασαφής. Μπορεί να είναι έγχρωμο όλο ο χάρτη, που σημαίνει ότι όλε οι χώρε δίνουν στοιχεία, αλλά αν πάτε στι περιφέρειε θα αρχίσετε να εντοπίζετε αδυναμίε. Επόμενη διαφάνεια. Ποια είναι η ε, φύση των στοιχείων ε, που δημοσιεύονται. Επιπλέον ε, ενημέρωση για τους δικαιούχους, αλλά πολύ λίγη και όχι και τόσο ενδιαφέρουσα θα έλεγα. Είναι η στοσελίδα και το τηλέφωνο του δικαιούχου στο 10% των περιπτώσεων που αναθεωρήσαμε. Ε, επιπλέον ε, προφορίες για τις δράσεις 40% ε, είναι η έδρα ας πούμε του δικαιούχου χωρισμένου για, για το καθεστώς και κάποια στοιχεία παρουσίασης και περιγραφής του έργου, του project και σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που έχουν εκταμιευθεί ποικίλει εκεί ο τρόπος με τον οποίο χορηγείται αυτή η οικονομική πληροφορία. Σε μερικέ περιπτώσει αναφέρεται μόνο το ποσό που έχει δεσμευτεί, η ανάληψη υποχρεώσεων δηλαδή, και σε άλλε περιπτώσει είναι οι πραγματικές πιστώσεις πληρωμών ή σε άλλες περιπτώσεις είναι μόνο ε, το μερίδιο που αναλογεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη χρηματοδότηση. Άλλοι αναφέρουν και το εθνικό ποσό. σε ό,τι αφορά τώρα την αξιοπιστία των στοιχείων και την ακρίβειά τους. Αυτό είναι στην απόλυτη ευκαιρία και τον έλεγχο των κρατών μελών και συγκεκριμένα των διαχειριστικών αρχών τους. για τα πραγματικώς καταβληθέντα ποσά, αυτό είναι από ορκωτού λογιστές και είναι προφανώς τα στοιχεία ακριβή. Αλλά για την ανάληψη υποχρεώσεων οι πηγέ είναι πιο ασαφεί. και εδώ έρχεται να προσθεθεί και ακόμα ένα πρόβλημα που έχει να κάνει ε, με το χειριστή που βάζει τα στοιχεία στο διαδίκτυο. Υπάρχει και ένα στοιχείο σφάλματος. Τώρα, χρησιμότητα βλέπετε ότι ο βαθμός, της λεπτομέρειας και τρόπος παρουσίασης στην ιστοσελίδα των στοιχείων διαφέρει πάρα πολύ από περιφέρεια σε περιφέρεια. Ιδιαίτερα το format, ε, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν PDF που δεν είναι πάρα πολύ φιλικό προς το χρήση. Δεν είναι πολύ εύκολο να βγουν τα στοιχεία εκεί και να τα χρησιμοποιήσουμε για περαιτέρω χρήση. Και έχουμε και διαφορές στις γλώσσες, στα νομίσματα, για χώρες που είναι εκτός ευρωζώνης. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνονται συγκρίσεις και πολλές φορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ανέφικτες. Δεν μπορεί να γίνει ε, συγκέντρωση των στοιχείων, aggregation των στατιστικών δηλαδή, ε, για να μην πω και για χρονοσύρες. Δηλαδή, γενικά, το θέμα ποιο είναι αυτό. Δεν είναι ε, ότι δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν εφαρμόζουν όσα τους ζητάμε τα κράτη-μέλη. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και στο περιεχόμενο και στον τρόπο με τον οποίο στέλνουν τα στοιχεία που δεν μπορούμε ούτε να τα ε, συνθέσουμε ούτε να τα συγκρίνουμε. Οπότε αμφισβητείται η χρησιμότητα των στοιχείων. Το πρώτο λοιπόν που κοιτάξαμε να δούμε γιατί σήμερα αυτό είναι ε, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια. Είναι τόσο διαφορετικά τα στοιχεία, δηλαδή τόσο πολύ ποικίλουν. Και ποιος είναι ο λόγος. Ένας από τους λόγους είναι ότι είναι πολλές επισημίες ως προς τα ελάχιστα στοιχεία. Τι είναι οι δικαιούχοι, τι είναι τα δημόσια ε, κονδύλια που δίνονται στις δράσεις. Με διαφορετικό τρόπο ερμηνεύονται αυτές οι έννοιες από κράτος σε κράτος και από περιφέρεια σε περιφέρεια. Τούτου λεχθέντος, ακόμα και αν είναι πλήρως εναρμονισμένα τα στοιχεία και αρμονική η κατανόηση του ορισμού, τι είναι δικαιούχος και τι είναι δημόσια κονδύλια, Παρ' όλα αυτά δεν αρκούν αυτά ως ελάχιστα στοιχεία. Είναι πολύ λίγα τα στοιχεία αυτά τα τρία. Να είναι χρήσιμα αυτά. Ως αντιπαράδειγμα, είδαμε στη Φιλανδία και την Πολανδία, η Πολωνία κυρίως, συγγνώμη, προγράμματα πολύ φιλόδοξα για δημοσίευση στοιχείων που έδιναν προφορίες για τους δικαιούχους και για τη λήψη των αποφάσεων για το ποια έργα χρηματοδοτούνται. και διάφορα κριτήρια που επιτρέπουν την έρευνα, ιδιαίτερα στην Πολωνία. Υπάρχει χάρτη για το σε ποιε περιφέρειε πηγαίνουν τα κονδύλια. Πολύ φιλικό προ το χρήστη, ε, τρόπο παρουσίαση είναι αυτό για του δικαιούχου. Το τελευταίο που έχει να κάνει με την πρωτοβουλία την ίδια είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια η ορατότητα του, της υποκείμενης λογικής, δηλαδή πώς είναι στημένο το, το σύστημα ολόκληρο. Οι διαχειριστικές ε, ε, αρχές προσπαθούν, αγωνίζονται να βρουν προφορίες που να μπορούν να αξιοποιήσουν, να τους χρησιμεύσει, να τους χρησιμεύσει γιατί. Ε, η δημοσιοποίηση των στοιχείων θα πρέπει να χρησιμεύει σε κάτι. Να δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα επικοινωνίας κάθε έργου η δημοσιοποίηση των δικαιούχων έχει στόχο να δίνει ενημέρωση για το τι χρειάζονται οι, δικαιούχοι, οι μελλοντικοί δικαιούχοι να γνωρίζουν για να συμμετέχουν και εκείνοι στο πρόβλημα. Δηλαδή δημοσιεύονται αυτά τα στοιχεία για να γίνεται το πρόγραμμα και το έργο πιο ελκυστικό. Γιατί προσπαθούν να συμπεριλάβουν και ε, νέα στοιχεία για την περιγραφή των έργων για τις βέλτιστες πρακτικές. Σε άλλες περιπτώσεις είδαμε τις διαχειριστικές αρχές να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για να ενημερώσουν για την έκβαση των προγραμμάτων, για την επιτυχία του προγράμματος. Δηλαδή θέλουν να δείξουν πού πηγαίνουν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι αποτέλεσμα έχουν αλλά εκεί επικρατεί αβεβαιότητα. Για ποιο λόγο να δημοσιεύονται οι κατάλογοι των δικαιούχων. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε τι στόχο εξυπηρετούμε κάθε φορά που δεν είναι σαφής. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συνδέονται με τα ίδια τα χαρακτηριστικά του συστήματος στη συνυπευθυνότητα, σε μεικτή διαχείριση. Η ενημέρωση για τους δικαιούχους γίνεται από τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν, εξορισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιορισμένο περιθώριο λιγμών. Αυτό κανονικά θα έδινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μεγαλύτερο καθοδηγητικό λόγο, μια που δεν έχει ρυθμιστικό. Αλλά ακριβώς ο καθοδηγητικός ρόλος λείπει. Και πώς εξηγείτε; θα σας πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ένας ογκόληθος. Από τη μια έχουμε το γραφείο του Αντιπροέδρου που άρχισε την πρωτοβουλία αυτή και τη λάνσαρε, αλλά από την άλλη έχουμε και τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι Γενική Διεύθυνση για την Περιφέρεια και Γενική Διεύθυνση ε, για την απασχόληση που εφαρμόζουν. Αν υπήρχε μεγάλη πολιτική βούληση στην αρχή που υπήρχε σε επίπεδο επιτρόπου για τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη, τη λογοδοσία κτλ. Αυτό δεν ε, υιοθετήθηκε απαραίτητο και από τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις που μπορεί να είχαν τις δικές τους προτεραιότητες και το δικό τους ε, έτσι, πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται αυτά τα δύο. Και τέλος, κοιτάξαμε τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Πολύ σύντομα σας αναφέρω μερικά στοιχεία, γιατί δεν ήταν καθοριστικά νομίζω στην εξήγηση ε, του κατά πόσο πέτυχε η ε, πρωτοβουλία αυτή. Το νομικό πλαίσιο δεν είναι εμπόδιο για τη σωστή εφαρμογή των απαιτήσεων. Το αντίθετο μάλιστα. Στη Φιλανδία για παράδειγμα ήταν ακόμα πιο ευνοϊκό. Πριν έρθει αυτή η πρωτοβουλία και η πρωτοβουλία ήρθε να αποτελέσει μάλλον επικάλυψη. Στη συνέχεια, το θεσμικό οικοδόμημα κάθε χώρα για τη διαχείριση των ε, διαρθρωτικών ταμείων, αν είναι κεντρικό ή αποκεντρωμένο, και πάλι δεν εμποδίζει, ούτε είναι εξήγηση. Κάποια τεχνικά στοιχεία είναι πιο σημαντικά για τη συλλογή του στοιχείου. Αυτό έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα τη διοικητική μηχανή να ανταπεξέρχεται στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα στι περιφέρειες. Αυτό είναι το θέμα τη Ιταλία. Ορισμένε περιφερειέ δεν είναι σε θέση να δημοσιεύουν τα στοιχεία αυτά διότι δεν έχουν τη διοικητική δυνατότητα να το κάνουν αυτό όταν είναι τεχνικά δύσκολο το πρόβλημα. Βέβαια έχουμε και πολιτικούς παράγοντες, ακόμα και πολιτιστικούς παράγοντες. Αλλά είναι μάλλον αποσπασματικά αυτά. Στην Πολωνία και στην Ισπανία. Για παράδειγμα στην Πολωνία δεν θέλουν να ε, δημοσιεύουν το όνομα των δικαιούχων για να αποφεύγονται αντιγραφές και δυσάρεστες συνέπειες. Συμπεράσματα. Ε, ε, κάθε χώρα δεν εφαρμόζει το πρόγραμμα με την πρωτοβουλία αυτή με τον ίδιο τρόπο. Αυτό έχει να κάνει με τη διοίκηση της χώρας με τον τρόπο τον οποίο έχει στηθεί η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Οι ελάχιστε απαιτήσει είναι ασαφείς, αμφίσιμες και, ε, εν πάση περιπτώσει, ανεπαρκείς. Και υπάρχει και ένα βαθύτερο πρόβλημα. Ο στόχος είναι συγκεχημένος ως προς την ε, ερμηνεία που δίνουν ε, τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες αυτό. Και έχουμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Από την αρχή ο στόχος ήταν πολιτικός και κατέληξε να είναι διοικητική ερμηνεία και ε, υπάρχει μια σύγχυση τώρα. Είναι πολιτικό αυτό που θέλουμε, είναι διοικητικό. Έχει επικρατήσει η διοικητική διάσταση της πολιτικής και την έχει επισκιάσει. Και ε, αυτό το σύστημα συν ε, διαχείρισης έχει και τα όρια του. Περνώ τώρα στις συστάσεις. είναι σε τρία επίπεδα. Πρώτο, σε πολιτικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Να επανέλθουμε στην αρχική επιθυμία και στον αρχικό σκοπό του Επιτρόπου κάλας. Να γίνεται από τους πολίτες ο κοινωνικός έλεγχος. Αυτή είναι η πολιτική προτεραιότητα. Για παράδειγμα, το κοινό θα πρέπει να γνωρίζει σε ένα συγκεκριμένο κλάδο εάν οι διαρθρωτικοί πόροι πηγαίνουν στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ας πούμε, στην Ήπεθρο. Ή αντίστοιχα, αν πηγαίνουν σε μεγάλους ομίλους ε, που εδρεύουν στις μεγάλες πόλεις. Ή ένας πολωνός αγρότης να ξέρει πόσα κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία πηγαίνουν στην περιφέρειά του και πόσα έχουν εκταμιεύσει οι αρμόδιες αρχές. Ή εγώ από περιέργεια, ας πούμε, θα θέλω να ξέρω στη γειτονιά μου ποιος πήρε κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία ή μια οργάνωση όπως αυτές που περιέγραψε ο κύριος Πρίτο να θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Αυτό δεν έχει να κάνει με την αξιολόγηση της πολιτικής. Συνδέεται με ένα, αλλά δεν ταυτίζεται. Ε, ούτε έχει να κάνει με το να ενημερώσει τους ε, ενδεχομένους δικαιούχους για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ταμεία. Ούτε με τον οικονομικό έλεγχο έχει να κάνει. Πάλι συνδέεται, αλλά δεν ταυτίζεται ακριβώς. Η δημοσίευση των δικαιούχων έχει στενή σχέση, αλλά και πάλι διαφορετική από άλλες δράσεις που είναι η επικοινωνία, ο έλεγχος. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι διαστάσεις που αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοενισχύονται και βοηθούν για τη διαφάνεια, αλλά είναι διαφορετική μεταξύ τους και θα πρέπει να έχουν και διαφορετική μεταχείριση. Δηλαδή, με το να δημοσιεύει απλώ ένα κατάλογο δικαιούχων, δεν καλύπτει όλου αυτού τους στόχου. Τώρα, δεν θα πρέπει να είμαστε στι ελάχιστες απαιτήσει, αλλά να έχουμε μια μαξιμαλιστική προσέγγιση. Τα κράτη-μέλη με μικρό περιφερειακό, περιθωριακό καλύτερα κόστος μπορούν να δημοσιεύουν περισσότερα στοιχεία και πιο χρήσιμα, εκτός από την απλή λίστα των δικαιούχων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καθοδηγεί περισσότερο, να θέτει το πλαίσιο, να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες όταν είναι πάρα πολύ ασθενής η κρατική μηχανή. Κυρώσεις. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό με το παρόν θεσμικό πλαίσιο. Θα ήταν καλύτερο να ποντάρουμε στην ήπια προσέγγιση που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα στο βαθμό που υπάρχει πραγματικός κοινωνικός έλεγχος. Και αυτό και πάλι έχει να κάνει και εξαρτάται από τη χρησιμότητα των στοιχείων. Τώρα, να περάσω στις πρακτικές βελτιώσεις. Θα πρέπει να μπουν και άλλα στοιχεία. Η έδρα, κοινωνικοί παράγοντες, ε, το μέγεθος ε, του έργου και με συγκεκριμένη ονοματολογία, ποιοι συμμετέχουν εκεί, με ποια υποστήριξη, από ποιο πρόγραμμα, ποιο ταμείο. Επίσης, αυτό ως προς την ουσία, ως προς τον τύπο τώρα, τον τρόπο με τον οποίο ε, παρουσιάζεται, ένα φόρμα με ενία ας πούμε γλώσσα, νόμισμα, υποστήριξη και για το Φεντέρ και αυτό και για το Κοινωνικό Ταμείο. Για να μπορούν να ε, ε, συναθρίζονται, να συνδυάζονται, να συνθέτουν τα στοιχεία, να συντίθενται μάλλον και να έχουμε και συγκρίσιμα στοιχεία. Για να μπορέσει η πρωτοβουλία αυτή να είναι πραγματικά πανευρωπαϊκή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι. Γι' αυτό ελπίζω να βοηθήσει για την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο και έμεσα. Γιατί είναι πραγματική φιλοδοξία αυτή και αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για αυτήν την ομιλία σας και τώρα να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένα στην κυρία Κατερίνα Ματερνόβα, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια για την Ανάπτυξη, τον Συντονισμό και την Κοινοποίηση της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκείνη θα μας παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής, ιδιαίτερως την ε, μελέτη στην οποία αναφέρθηκε και η κυρία Πελεγκρίν. Πρέπει Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την ενδιαφερουσότατη εκδήλωση. Μια στιγμή όμως να μαζέψω τα χαρτιά μου εδώ γιατί κρατούσα σημειώσεις. Όπως άκουγα την παρουσίαση της κυρίας Πελεγρίνου. Όπως ξέρουν ήδη οι συνεργάτες μου, δεν θα μιλήσω από τα χαρτιά όμως, αλλά από στήθους. Α, να, να. Λοιπόν, καταρχάς, γενικά ως άνθρωπος που μπήκε στην Επιτροπή λίγους μήνες πριν αρχίσει η πρωτοβουλία διαφάνειας του Επιτρόπου Κάλας, Πρέπει να σας πω ότι ο Γενικός Διευθυντής ενθουσιάστηκε από αυτή την ιδέα και ο τότε Αντιπρόεδρος απογοητεύτηκε κάπως γιατί οι υπόλοιπε υπηρεσίες δεν έδειξαν τον ίδιο ενθουσιασμό. Εγώ είμαι αγωνίστρια υπέρ της ελευθεροτυπίας ήδη από τη Βουλγαρία και γι' αυτό εγώ χάρηκα ιδιαίτερα από την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι όπως και στη Γενική Διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ενός τρίτου του προϋπολογισμού. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο πολίτης πού πηγαίνουν τα χρήματα. Και όχι μόνο για τη διαφάνεια αλλά και για άλλα θέματα πολλοί πολίτες θεωρούν ότι δεν συμμετέχουν αρκετά Ό,τι δείκτες και να συλλέξουμε δεν αρκεί αυτό. Δεν το λέω για δικαιολογία, όχι είναι μια εξήγηση. Θα συλλέξουμε δείκτες και άλλους. Στο νέο πλαίσιο σίγουρα θα το κάνουμε. Διότι η πρωτοβουλία διαφάνειας ήρθε μετά από τον καθορισμό των δημοσιονομικών προοπτικών αλλά πάντως στην περίοδο 7 με 13 γνωρίσαμε την πρώτη φορά από τον προϋπολογισμό και συμφωνώ εδώ με το σχόλιο της κυρίας ότι, ότι δηλαδή για πρώτη φορά λέω στον προϋπολογισμό φάνηκε ότι μερικές χώρες μέλη ακολουθούν το γράμμα αλλά όχι το πνεύμα της πρωτοβουλίας άλλες όμως αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα, υποδείγματα θα έλεγα, Λιθουανία, Ουγγαρία, Φιλανδία, Γαλλία, που πήραν τα ελάχιστα αυτά που προέβλεπε το νομοσχέδιο και τα προσήφξησαν για να υπάρχει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα και άλλα και νομίζω ότι το επόμενο βήμα θα είναι ακριβώς αυτό να είναι σε πανενοσιακό επίπεδο τα στοιχεία συγκρίσιμα και και, και λέγω είναι πάντοτε δύσκολο να μεταφερθούν συστήματα από το εθνικό στο ενωσιακό επίπεδο αλλά σίγουρα θα το θα το προσπαθήσουμε αυτό, θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι στα πλαίσια της δομής μας του shared management όπως λέμε εξαρτώμεθα από την καλή θέληση δυστυχώς των, καλών, των χωρών μελών και περιφερειών. Προσπαθήσαμε να προμηθεύσουμε, να χορηγήσουμε, να δημιουργήσουμε ελάχιστα κοινά πρότυπα και μετά κάναμε και δύο πρόσθετα βήματα τη δημιουργία μίας θηρίδας ίντερνετ, θύρας μάλλον, ή πύλης, για να υπάρξει μεγαλύτερη πρόσβαση από τους χρήστες και σε καταλληλότερη μορφή. Και μετά δημιουργήσαμε ένα δίκτυο 250 υπαλλήλων επικοινωνίας που συνεδριάζουν ετησίως και ανταλλάσσουν τις εμπειρίες των είναι λίγο σαν μετεκπαίδευση αλλά ιδιαίτερα ανταλλαγή βελτίστων όπως λέμε. Λοιπόν, Εμεί εδώ στην πολιτική συνοχή δεν θεωρούμε ότι ανταποκρινόμαστε μόνο στο τελευταίο στοιχείο της πρωτοβουλίας διαφάνειας, δηλαδή τους ε, από τα ταμεία, αλλά θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχής αφορά και άλλες πτυχές της γενικότερης διαφάνειας, όπως τη διαδικασία διαβούλευσης. Τώρα συζητάμε πρωτοβουλίες και συστάσεις ε, όπως το Using Your Voice Europe. Επίσης θεωρούμε ότι ότι είμαστε σε θέση να χορηγήσουμε πληροφορίες για τους δυνητικούς χρήστες και ε, αυτό θα θέλαμε να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Μέρος της διαδικασίας αυτής είναι αυτή η κίνηση για απλοποίηση και ο κατακαιρματισμός των προγραμμάτων και των πολιτικών με την πιθανή τους ή τις πιθανές τους επικαλύψεις από διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα που καταλήγουν στον ίδιο αποδέκτη είναι τμήμα και αυτό της προσπάθειάς μας αυτή. Δεν ξέρω αν θα λυθεί εύκολα αλλά σίγουρα τουλάχιστον μπορούμε να δώσουμε τις πληροφορίες με πιο συνεπή και συνεκτικό τρόπο και σε συνεννόηση και με άλλους βέβαια αρμόδιους ώστε τουλάχιστον στο μέλλον η πληροφόρηση να χορηγείται με τρόπο φιλικότερο προς τον χρήστη και την χρήστρια Το ξαναλέω ότι δεν είναι δικαιολογία αλλά εξήγηση. Αυτή η δομή του shared management είναι τέτοια ώστε, ώστε λέγω ο ευκολότερος τρόπος να φτάσει κανείς να πετύχει κανείς ορισμένα στόχους επιτυχάνεται μόνον αφού καθοριστεί οι πολυε... το... στούν οι δημοσιονομικές προοπτικές και αφού εγκριθούν αυτές είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να αλλάξουν οι κανόνες και να γίνουν αυστηρότεροι. Εδώ λοιπόν εξαρτόμαστε ε! από την καλή θέληση και το ενδιαφέρον των χαρών μελών. Το σχόλιο σας λοιπόν κυρία Πελεγρίν για, την, για τον παράγοντα της καλής πολιτικής θέλησης είναι ακριβώς αυτό που ισχύει και που εξηγεί τις μεγάλες διαφορές στη στάση των χωρών μελών, πόσο θέλουν δηλαδή, πώς είναι η θέλησή τους. Ξέρετε ίσως ότι ότι η Λιθουανία πήρε βραβεία τελευταίως, βραβείο διαφανίας γιατί χορήγησε πληροφορίες προς τους ωφελουμένους και χρήστες και χρήστριες και οφελούμενες Και απ' την άλλη πλευρά βέβαια δεν έχουν όλη την ίδια στάση, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και εμείς θέλουμε, θέλουμε να, στο μέλλον να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια ήδη από το επίπεδο της συγγραφής των νομοσχεδίων, της σύνταξης των νομοσχεδίων. Ε? Να γίνουν δηλαδή μελέτες κλπ. Παράδειγμα, δεν είναι βέβαια για διαφάνεια αλλά από τους ωφελουμένους, αλλά τουλάχιστον προς τους δυνητικούς ωφελουμένους ή πλασματικούς ωφελούμενους. Οι διαχειριστικές αρχές θα μπορούσαν να γνωστοποιήσουν, να γνωστοποιούν αν υπάρχουν ευρωπαϊκά ταμεία για κάποιο πρόγραμμα, γιατί σε μερικές χώρες είναι πολύ δύσκολο να γνωστοποιούνται όλα αυτά. Δεν γνωστοποιούνται. γνωστοποιούνται. Και δεν γνωρίζουν επομένως οι πολίτες και οι πολίτησες ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε μια Ευρώπη των 27 και η τελευταία μελέτη δείχνει ότι υπήρξε μεν κάποια πρόοδος αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλές και άλλες για να τα πάρουμε υπόψη μας και εξάντε και εξπόστο όπως εξάλλου πρέπει. Επομένως ήδη από τη φάση της σύνταξης των νομοσχεδίων πρέπει να είναι όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για τη συνεισφορά της και τώρα να ακούσουμε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μόρτεν Λέβισον, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που θα μας μιλήσει συγκεκριμένα για τη σχέση μεταξύ διαφάνεια και ευθύνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή να του προπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου για αυτή την ενδιαφέρουσα και σημαντική ακρόαση που οργάνωσε για τη διαφάνεια στα διαφορετικά ταμεία. Το πληροφορήθηκα πριν από δύο μέρε περίπου και ήταν πολύ σημαντικό που μπόρεσα να ακούσω όλε αυτέ τι συνεισφορέ και χαίρομαι που προσκεκλήθη ω ε, ομιλητή εδώ, ω μέλο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην απόφαση τη 19η Φεβρουαρίου 2008 για τη διαφάνεια στα δημοσιονομικά ζητήματα, το Ευρωκοινοβούλιο έχει ήδη τονίσει ότι η διαφάνεια συνεισφέρει στην ενίσχυση των αρχών τη δημοκρατία και του σεβασμού των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η θέση αυτή πρόσφατα επιβεβαιώθηκε από το Κοινοβούλιο στην απόφαση της 15ης Ιουνίου 2010 περί διαφάνειας στην ε, περιφερειακή πολιτική. Έχει προσαρτηθεί και στο φάκελο μια απόφαση αυτή. Στο επίπεδο των διευθυντικών ε, ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των παρεμβάσεων τους, η διαφάνεια για μας σημαίνει ότι διασφαλίζουμε πρώτα απ' όλα μια σαφή κατανόηση μεταξύ των δυνάμει ε, δικαιούχων για τον τρόπο που παρέχεται η ευρωπαϊκή στήριξη, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε αυτή τη στήριξη και έπειτα πρέπει να διασφαλίζει την παροχή στους Ευρωπαίους πολίτες και ενδιαφερομένους αξιόπιστων και ε, εύστοχων πληροφοριών για το πώς έχουν δαπανηθεί τα κονδύλια. Και έπειτα να είναι διαθέσιμες αξιόπιστες και στοιχετικές ε, πληροφορίες για τις και τα αποτελέσματα των ε, παρεμβάσεων των διευθυντικών ταμείων, επιτρέποντας τους Ευρωπαίους ενδιαφερομένους να αποτιμήσουν την αποτελεσματικότητα και την ε, οικονομία που επιτυγχάνουν οι παρεμβάσεις αυτές και έπειτα η λογοδοσία όσων έχουν επενδυθεί με την ευθύνη διαχείρισης των δημοσίων κονδυλίων. Η κατάρτιση καταλόγων των δικαιούχων της ευρωπαϊκής στήριξης ε, ανταποκρίνεται σε αυτές τις ε, ανησυχίες και μέρημνες. Το να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για πληροφόρηση, σεβασμού του ιδιωτικού βίου και του επιχειρηματικού απορρίτου είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Εγώ ίδιος, όντας ελεγκτής, δεν θα σας πω ποια ακριβώς είναι η σωστή ισορροπία ή τι είδους πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στους Ευρωπαίους πολίτε. Απλώ καταγράφω την απόφαση του Επινοβουλίου τη 15η Ιουνίου 2010. Περισσότερο θα ήθελα να σταθώ στι αδυναμίε που έχει παρατηρήσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με τη διαφάνεια και τι συστάσει που έχουμε εκδώσει σχετικά. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να επικεντρωθώ στην διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία για την επικαιρότητα των πληροφοριών, που είναι τρεις βασικές πτυχές, τις οποίες θα πρέπει να δούμε προκειμένου να επιτύχουμε πραγματική διαφάνεια και λογοδοσία. Τα διευθυντικά ταμεία και οι δραστηριότητέ του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκε εξαιτία του υψηλού αριθμού συγχραματοδοτουμένων προγραμμάτων και επειδή είναι μεγάλη η ποικιλία του είδους και της μορφής των προγραμμάτων. Αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, ε, τμήματα σιδηροδρομικών ε, συνδέσεων, ε, μονάδες επεξεργασίας υδάτων, κεφάλαια κινδύνου, τουριστικές υποδομές και ούτω καθεξής. Το φάσμα των δικαιούχων είναι μεγάλο και μπλέκονται δημόσιοι φορείς, εθνικοί τοπικές περιφερειακές αρχές, ε, δημοτικές αρχές, πανεπιστήμια και το καθεξής. Και ιδιώτες, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώσεις που παρέχουν εκπαίδευση, ή ιδιώτες και ούτω καθεξής. Ε, το να έχουμε επίκαιρες και εύστοχες πληροφορίες ε, σε σχέση με το κόστος και τα αποτελέσματα είναι κάτι που ε, διαρκώς επιζητά το ελεγκτικό συνέδριο στις αιτήσει και ειδικέ εκθέσεις, του. Τώρα για την νομιμότητα και τη συστηματικότητα των δράσεων των διαφορετικών ταμείων, αυτό είναι μέρος της αξιοπιστίας των πληροφοριών. Εδώ το ε, συνέδριο σημείωσε στις αιτήσει εκθέσεις του ότι τα σφάλματα συνήθως προέρχονται πρώτον από ε, αιτήσει αξιώσεις που δεν είναι επιλέξιμες από πλευράς δικαιούχων ε, δεν είναι επιλέξιμες ε, γιατί το κόστος δεν σχετίζεται με το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή δεν μπορεί να καλυφθεί από την περίοδο προγραμματισμού. Επιτά υπάρχει μια τάση υπέρμετρης δήλωσης των επιλέξιμο, το επιλέξιμο κόστος. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ασφάλματα αυτά έχουν να κάνουν ε, με προσωπικό που έχει υπερεκτιμηθεί ή με υπερβολικά εκτιμημένα κόστη. Και δεν έχουν σωστά αφαιρεθεί, δεν έχει σωστά γίνει η αναλογία εισοδημάτων και κόστους, εσόδων και κόστους. Ή η μη συμμόρφωση με τους κανόνες δημοσίων προμηθειών. Εδώ έχουμε ένα τομέα που κλασικά η διαφάνεια είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων της προμήθειας. Καθώς υπάρχουν ελλείψεις στα συστήματα ελέγχου και ο τελικός δικαιούχος πρέπει να εντοπίζεται. Ε, εντοπίζουμε έτσι και μια σημαντική πηγή σφαλμάτων. Το συνέδριο λοιπόν συστήνει στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των 100 μελών μια έγκαιρη μορφή συνεργασίας μεταξύ των αρχών διαχείρισης για το πρόγραμμα και αυτών που διαχειρίζονται το πρόγραμμα ώστε να εξοικειωθούν με, τα, με τους κινδύνους ε, σφάλματος και νομικής συμμόρφωσης. Επίσης, σωστή επιλογή και κατάρτιση του προσωπικού προκειμένου να προλαμβάνονται και να εντοπίζονται σφάλματα στις δηλώσεις κόστους των προγραμμάτων και στις διαδικασίες των δικαιούχων. Και επίσης αποτελεσματική επίβλεψη από την πλευρά της Επιτροπής και βασική έλεγχη στα κράτη-μέλη ε, βάσει της ανάλυσης κινδύνου των συστημάτων ελέγχου των διάφορων αρχών διαχείρισης. Ωστόσο το συνέδριο τόνισε ότι υπάρχει και ένα όριο στις βελτιώσεις που μπορούν να επιφερθούν στην εποπτεία και διαχείριση και επίβλεψη μάλλον και στον έλεγχο χωρίς να υπάρχει ανάγκη ε, ριζικής μεταρρύθμισης των υποκείμενων κανόνων και κανονισμών. Επειδή αυξάνεται ο αριθμό των ελέγχων και τα σφάλματα γίνονται λιγότερο συχνά, το κόστος των ελέγχων μπορεί κάποια στιγμή να αρχίσει να υπερβαίνει το όφελος του περαιτέρω περιορισμού των σφαλμάτων. Από την άλλη πρέπει να τονίσω ότι ίσως να υπάρχει ακόμη περιθώριο για βελτίωση ποιότητας και αποτελεσ... ποιότητα ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων ελέγχων. Έτσι λοιπόν ανάγκη για διαφάνεια υπάρχει, αλλά και στους ελέγχους και στο κόστος των ελέγχων και τις σχετικές τους πληροφορίες, ώστε να μπορούμε να αποτιμήσουμε πού είναι το σωστό σημείο ισορροπίας. Όπου δεν μπορεί να εξευρεθεί τέτοιου είδους ισορροπία, πρέπει είτε να υπάρξει μεταρρύθμιση, είτε να επανεξεταστούν τα προγράμματα και τα σχέδια υπό εξέταση. Μια δεύτερη σωματική πηγή σφαλμάτων έχει να κάνει με την πολυπλοκότητα των κανόνων επιλεξιμότητας και άλλες προποθέσει στις οποίες υπόκεινται οι δικαιούχοι. Η απλούστευση είναι ένας τρόπος να ενθαρρύνουμε τη διαφάνεια και θα πρέπει να παραμείνει μια από τι πρώτε μα προτεραιότητε. Οι κανόνε και οι κανονισμοί πρέπει να είναι σαφοί, να μπορούν να ερμηνευθούν, να εφαρμοστούν με απλό τρόπο και να ε, μειώνουν το επίπεδο κινδύνου καθώς και τα, το κόστος του ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να αποτιμηθούν οι συνέπειες της ποιότητας της δαπάνης. Επίσης το συνέδριο τόνισε ότι τα ε, εξή στοιχεία συνδέονται άμεσα με τη διαφάνεια και πρέπει να βελτιωθούν. Πρώτον, οι αποτιμήσεις που γίνονται στις ε, εκθέσεις ετήσιας δραστηριότητα και τις δηλώσεις των Γενικών Διευθυντών της Επιτροπής ως προς την αξιοπιστία των εσωτερικών ελέγχων για τομείς υψηλού κινδύνου. Και έπειτα, στην ποιότητα των δεδομένων που τα κράτη-μέλη απαιτούν του απαιτείται να παρέχουν ε, στην Επιτροπή ως προς τους δημοσιονομικές διορθώσεις και τους μηχανισμούς ανάκτησης. Ο δεύτερος βασικός τομέας ε, στον οποίο έλεγχο το συνεδριό μας είναι η αποτελεσματικότητα, η υποδοτικότητα και η οικονομία που επιτυγχάνουν οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ε, κλασικές ειδικές, στις ειδικές μας μάλλον εκθέσεις. Σε ό,τι αφορά τα κύρια προγράμματα, όπως έχει σημειώσει και το συνέδριο στην ειδική έκθεση 1-2008, υπάρχει ανάγκη για περισσότερο αποτελεσματική και συνεπή προκαταρκτική εξέταση, πρώτερη εξέταση των αιτήσεων για προγράμματα σε επίπεδο Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ορίσει ένα πολύ υψηλό ποσοστό κοινοτική συμβολή σε πολλές περιπτώσεις. Το συνέδριο συστήνει να ενταθούν οι προσπάθειες για να καταρτιστούν κανόνες προσαρμογής της ε, κοινοτική συμμετοχής κατά τρόπο συνεπή, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό διαφάνειας των ε, ευρωπαϊκών δαπανών. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες από την Επιτροπή για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και το αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί από το συνέδριο στους μελλοντικού του ελέγχους. Οι αδυναμίες πολλές φορές αφορούν την έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με τις επιδόσεις και αυτό βεβαίως υπονομεύει την λογοδοσία. Το συνέδριο έχει παρατηρήσει πολλές περιπτώσεις όπου οι στόχοι και οι σχετικοί δείκτες δεν έχουν οριστεί επαρκώς. Αυτό δεν επιτρέπει να καταμετρηθούν οι επιδόσεις του προγράμματος. Επίσης, όπου οι στόχοι και οι δείκτες έχουν οριστεί, παραμένουν πολλές περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες για το αποτέλεσμα και τον αντίκτυπο απουσιάζουν, είναι ανεπαρκείς ή δεν είναι αξιόπιστες. Αυτό έχει σημειωθεί και στην ειδική έκθεση 10-2006 σχετικά με την ε, exposed ε, αποτίμηση, την έκθεση 1-2007 για τις ενδιάμεσες διαδικασίες και επίσης την ειδική έκθεση, την πιο πρόσφατη 1 του 2008 για τα κύρια προγράμματα και την 17η του 2009 για την επαγγελματική κατάρτιση για τις γυναίκες και τις σχετικές δράσεις για τις γυναίκες μάλλον. Αυτές οι ελλείψεις δυσκολεύουν ε, την ε, αποτίμηση του κατά πόσον σωστά δαπανούνται τα κονδύλια και τους ελέγχους. Έτσι λοιπόν το συνέδριο σε σχέση με τα διαρθρωτικά ε, ταμεία πρέπει να συλλέγει πληροφορίε σε επίπεδο δικαιούχου για τα αποτελέσματα. Η έλλειψη πληροφοριών σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε σωστά σύνολα πληροφοριών για το τι έχει επιτευχθεί μέσω τη οικονομική βοήθεια των διευθυντικών ταμείων. Το όρο SMART σημαίνει συγκεκριμένο, μετρήσιμο, εφικτό, αξιόπιστο και επίκαιρο. Το, συνέδριο λοιπόν ε, πρότεινε οι στόχοι SMART και οι σχετικέ επιδόσει και οι δείκτε του να συλλέγονται και να διατίθενται με τρόπο συστηματικό. Ε, γενικότερα το συνέδριο συνέστησε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει κατά πόσον υπάρχει περιθώριο να επικεντρώνεται σε περισσότερα αποτελέσματα παρά ποσοτικά αποτελέσματα και αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί έμφαση βελτίωση της, της καλής διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών και έτσι θα ενισχυθεί και η διαφάνεια. Πρόεδρε, ε, κύριοι βουλευτές, ε, μέλη της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, κυρίες και κύριοι, ναι, έχει επιτευχθεί πρόοδος προς την ε, αύξηση της διαφάνειας, την διαχείριση των διευθυντικών ταμείων και προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και ενδιαφερομένων. Έτσι, η περισσότερη διαφάνεια θα ενισχύσει τη λογοδοσία όσων είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επιπλέον, περισσότερο διαφανεί πληροφορίε για την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την οικονομία που την χάνουν τα διευθυντικά ταμεία και οι δαπάνε του, θα μα οδηγήσουν και σε καλύτερο ορισμό τη συγκεκριμένη φύση και μορφή που θα χρειαστούν μελλοντικέ παρεμβάσει και για τι απαραίτητε βελτιώσει που θα χρειαστούμε για την οργάνωσή του. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά. Στη συζήτηση έχει ζητήσει το λόγο βεβαίω ο συνάδελφο Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μα λέτε. Θέλω να πω στην κυρία Πελεγκρίνο όμω ότι δεν μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που προσπαθεί να αλλάξει ως ιστορική πραγματικότητα. Ποια είναι η ιστορική πραγματικότητα. Καλά τα ξεκίνησε ο κύριος Κάλλας, αλλά δεν έγιναν νόμοι ζητήθηκε από την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια, που ήταν όμως ανακοίνωση, νομοθετική ε, εφαρμογή μετά από τροπολογίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πουθενά δεν προτάθηκαν αυτά που ζητούσαμε. Δημοσίευση των δικαιούχων. Τα ξέρω αυτά γιατί ήμουν και εγώ η ίδια ε, ε, στο δημοσιονομικό κανονισμό εισηγήτρια και εμείς το βάλαμε η ε, περιφερειακή πολιτική, τα διορθωτικά ταμεία, μετά ο προϋπολογισμός και μετά έκανε μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα γεωργικά. Έτσι για να αποκαταστήσουμε και την ιστορική αλήθεια. Και από την αρχή πήγε στραβά. Αυτή η ιστορία του ownership δεν το είχαν στενιστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν το είχαν κάνει κτήμα τους, το είχε προτείνει ο κύριο Κάλλα, αλλά νομοθετικά δεν το υλοποίησε. Ούτε ο ίδιο είχε τη δύναμη να το επιβάλλει νομοθετικά. Και μέχρι σήμερα υφιστάμεθα τι συνέπειε, γιατί στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να ορίσει τι θέλει να δημοσιεύεται. Το Κοινοβούλιο και εγώ ίδια έχω κάνει προτάσει και στο δημοσιονομικό κανονισμό και στι εκτελεστικέ διατάξει και εκ των υστέρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά δεν υιοθετήθηκαν. Δηλαδή σήμερα πάσχουμε από αυτό το πρόβλημα. Το έχουμε εντοπίσει ότι χρειαζόμαστε εναρμόνιση, αυτή τη δυνατότητα όμως δεν την αξιοποιήσαμε. Οπότε αγαπητή κυρία μου ε, Ματχτένοβα, δεν μας τα λέτε καλά ότι κάνουμε τεράστιες προσπάθειες και έχουμε τεράστια βούληση, αλλά τα κράτη-μέλη δεν βοηθάνε, γιατί βοηθάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν με ικανοποιούν καθόλου αυτά που μας είπατε, διότι πραγματικά λέμε ότι ο δρόμος προς την κόλαση, και αυτό το δρόμο έχετε πάρει, είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Και αν συνεχίσετε αυτή την ατραπό, άλλα δέκα χρόνια τα ίδια θα λέμε. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει προτάσεις εφικτές, δεν θα μπορούσαν να τις υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη και πάνε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ενιαία γλώσσα. Αγγλικά. Lingua franca. Ενιαίες τιμές. Ενιαίες ρυθμίσεις. Γιατί θέλουμε να δημοσιεύονται οι αποδέκτες. Καλή η διαφάνεια, αλλά να έχει και ένα στόχο. Όχι για τη διαφάνεια, δεν είναι αυτό ο σκοπός. Θα πρέπει να δούμε αν έχουμε καλύψει τον πολιτικό μα στόχο. Α πούμε, τα διορθωτικά ταμεία, τα γεωργικά ταμεία εξυπηρετούν το στόχο που έχει η πολιτική μα. Γι' αυτό τα μετράμε, γι' αυτό θέλουμε να δημοσιεύονται, για να είναι και συγκρίσιμα. Πιάνουν τόπο τα λεφτά μα. Τώρα έχουμε ένα νεκροταφείο στοιχείων. Μα έχουν κατακλείσει. Τι να τα κάνουμε όμως αυτά, να τα αξιοποιήσουμε πολιτικά. Και θα σκεφτόμουν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο συνομιλητή. Πολύ ωραία δουλειά για την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Θεμάτων. Να καθίσει, να τα αναλύσει, να εξηγήσει ποιο παίρνει τα λεφτά στα κρατημέλη, τι τα κάνει και αν φτάνουμε στους στόχους μας. Γιατί αυτά που ακούω πραγματικά ανατριχιάζω. Το πέμπτο, ας πούμε, πολυτελές ξενοδοχείο σε ένα σλοβενικό χωριό. Μα μου λένε ποιοι ε, χρηματοδοτούν αυτές τις ανοησίες. Μέχρι σχολεία χτίζουμε. Μα αυτό είναι στην επικουρικότητα, στα κράτη-μέλη. Τέτοια πράγματα χρειαζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μου, μου έχει σηκωθεί η τρίχα από αυτά που ακούω. Να μην τα λέει μόνο η κυρία Πελεγκρίν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει. Με ένα κατάλογο ε, για τις χειρότερες επιδόσεις ας πούμε. Και τι θα τους κάνουμε αυτούς. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στο νέο κανονισμό, στη νέα ρύθμιση και είναι και συναπόφαση τώρα, να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συνδέουμε τη χρηματοδότηση και με τη δημοσίευση των στοιχείων για το πώς τα δαπανούμε τα κονδύλια αυτά και θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα αυτό που μας είπαν οι κύριοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δικαιούχος υποχρεούται τέσσερις φορές το χρόνο να τα δηλώνει αυτά και μιλάμε για χιλιάδες δικαιούχους. Εμείς τι συμπεράσματα θα βγάλουμε από τις δημοσίευσεις λοιπόν. Αυτό θα ήταν ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί δεν βελτιώνεται τα πράγματα. Γιατί δεν θέλετε να σας εξοδοτήσουν για τις εκτελεστικές ρυθμίσεις, τις οποίες μπορείτε να προσαρμόζετε. Μην νομίζετε ότι θα κάνετε ένα κανονισμό για 7 χρόνια χωρίς καμία τροποποίηση. Πρώτη φορά ακούω τέτοια πράγματα. Έχω ανατριχιάσει. Αν είχαμε και καλή βούληση και βούληση σκέτο να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά τα πράγματα, θα πήγαιναν πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Μπαλτσίτης. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους μας για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας χορήγησαν και γιατί μας ανέφεραν και την εμπειρία άλλων χωρών και περιφερειών όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ακούσαμε πολλά θετικά σχόλια για τη Λιθουανία και εγώ ήμουν από εκείνου που από τους προτεργάτες της δημιουργίας της ιστοσελίδας που αναφέρθηκε στις παρουσιάσεις. Μετά από τότε άλλαξαν πολλές κυβερνήσεις και δεν ήξερα καν ότι είχε πάρει αυτό το βραβείο διαφανείας η Λιθουανία. Συμφωνώ με τον συνάδελφο που μίλησε πριν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει όμως ως προς τη στάση των χωρών μελών. Όλα αλλάζουν, πάντα ρί και η, η ζωή αλλάζει. 300 δισεκατομμύρια ευρώ δίνονται στα κράτη-μέλη για τη βελτίωση, λέει, της ανταγωνιστικότητάς τους. Αλλά η Κομισιόν δεν καθορίζει ακριβώς ποιες είναι οι ευθύνες ποιον. Εγώ έχω σημειώσει πράγματα που είπε σήμερα η κυρία Πελεγκρίν Δηλαδή, πώς μπορεί να αναμένει κανείς ότι τα κράτη-μέλη θα χορηγήσουν αξιόπιστες πληροφορίες, μας είπε. Και η κυρία Ματέρνοβα, εκπροσωπώντας την Κομισιόν, μας είπε σήμερα η πληροφόρηση εξαρτάται από την καλή θέληση των χωρών μελών. Αυτά είναι δύο βασικά στοιχεία που πρέπει να τονίσουμε. Θυμάμαι την εποχή που τα κράτη-μέλη έπρεπε όντως να δημιουργήσουν μόνα τους τα συστήματά τους. Το είχα κάνει και εγώ στη Λιθουανία, μας είχαν αφήσει μόνους, κατάμονους. Δεν μπορούσαμε βέβαια να τα κάνουμε όλα από το μηδέν γιατί κάθε χώρα είχε κάποια, κάποια ήθη και συνήθειες για τη συλλογή των πληροφοριών. Άλλοι μας είπαν σήμερα ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τους πολίτες και ιδιαίτερα το προσωπικό των Υπουργείων. Το θέμα το ξέρω ότι είναι λεπτό, το ξέρω, αλλά πρέπει να σας πω ότι σε πολύ, σύντομα θα χρειαστεί να πάρουμε αποφάσεις. Και εδώ πρέπει να βασιστούμε νομίζω στην εμπειρία των ήπα η Κομισιόν δηλαδή να ορίσει έναν υπεύθυνο για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων για τη διαφάνειά τους. Διότι σήμερα ζητούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Απλοποίηση των κανόνων από τη μία και από την άλλη απαιτούμε από τα κράτη-μέλη να απορροφούν σωστά 100% τα κονδύλια. Μα ποιος αρχηγός κράτους μπορεί να αρχίσει η απλοποίηση των κανόνων άμα γνωρίζει ότι θα θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνο για το παραμικρότερο λάθος. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει εδώ να αναλάβει τις ευθύνες της. Όσοι οι καταλληλότεροι να αναλάβουν τις ευθύνες αυτές πρέπει να οριστούν, να διοριστούν και αυτοί να κάνουν την απολοποίηση στα κράτη-μέλη. Τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν σήμερα για τις Ηνωμένε Πολιτείε ήταν νομίζω πολύ χρήσιμα στο μέλλον. Θα έπρεπε όλες αυτές οι διαδικασίες να συνδέονται και με το κοινό. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αναπνεύσουμε. οι κυβερνήσεις δηλαδή και οι υπεύθυνοι γενικότερα. Εγώ δεν έχω ερώτηση να θέσω αλλά ένα σχόλιο να κάνω ήθελα. Θα κάνω ό,τι μπορώ και εγώ ώστε να πιέσω την Κομισιόν να αναλάβει τις ευθύνες της και στα 27 κράτη-μέλη. Αφού δεν μιλάμε για το ρυθμό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ξέρω ότι τελειώνει η προγραμματική περίοδος, πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι μερικές χώρες μέλη δεν είναι σε θέση να τα απορροφήσουν 100%. Δεν είναι σε θέση. Ευχαριστώ κύριο Στάς. Ehm, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακρόαση είναι εδώ για να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον. Και όπως είπε ο προλαλή σα, σήμερα το πρωί ακούσαμε νέα πράγματα και μάθαμε πώς λειτουργούν αυτά στις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν μ' αρέσουν οι μονόλογοι. Και μια φορά είχαμε μονολόγους στο παρελθόν, ο καθένα ερχόταν εδώ, έλεγε το πείματάκι του, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον κτλ. Ε, αλλά οι τρεις τελευταίοι, κύριε Λέβισον, εσείς μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, η κυρία ε, Ματερνόβα που είναι από τους πιο υψηλόβαθμους υπαλλήλου στη Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειακών Θεμάτων και στην κυρία Πελεκρίν, ε, ακαδημαϊκό. Εσείς τι μάθατε, θέλω να σας ρωτήσω, από τον κύριο Μπρίτο και τον κύριο Ντέβανη, αυτό που μας είπαν το πρωί, που να μας λέτε ότι ορίστε, αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλουμε να το μελετήσουμε περισσότερο και να το σημειώσουμε για μελλοντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Grazie, ε, ευχαριστώ, κύριε Σόνεργκάρτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και μένα μου άρεσαν αυτά που άκουσα και σας ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής, που νομίζω είναι σχετικό. Εκτός από την έλλειψη της πολιτικής βούλησης, τι εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει ένα σύστημα όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, από οποιοδήποτε σημείο της χώρας να μπαίνει κανείς σε μια κεντρική βάση δεδομένων και να ψάχνει ποιο πήρε και ποια κονδύλια. Τι μας ε, εμποδίζει να το κάνουμε αυτό, μπορείτε να μου εξηγήσετε σας παρακαλώ πολύ. Και θέλω να θυμίσω ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι θεμελιώδες δικαίωμα, δεν το γράφει η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να είσαι δικαιούχος και αποδέξεις βοήθειας. Και ένα από τους όρου αυτούς είναι να βοηθάς και να ενημερώνεις συγκεκριμένα μια τέτοια βάση δεδομένων. Θα έλεγα λοιπόν στους τρεις τελευταίους ομιλητές, πέρα από την πολιτική βούληση λοιπόν, τι εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει αντίστοιχο σύστημα με των Ηνωμένων Πολιτειών. Κύριος Χατζημαρκάκης παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, και είναι ερώτηση αυτή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να συμπληρώσω αυτά που είπε η κυρία Γκρέσλε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να απορρίπτει την ευθύνη ε, για την ακρίβεια των στοιχείων. Εντάξει, το σημειώνουμε. Αλλά δεν είμαστε πλέον πρόθυμοι να το δεχθούμε. Εγώ δεν θα είμαι τόσο οξύ όπω η κυρία Γκρέσλε, αλλά επί τη ουσία εξίσου σαφή. Γιατί να δεχόμαστε εμεί ότι η ακρίβεια δεν είναι δεδομένη. Διότι και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία ενός νέου κράτους μέλους. Δεν βοηθήθηκε κανείς. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε τα κράτη-μέλη να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνδέσει τη χρηματοδότηση με την τήρηση κανόνων, τότε θα συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Και ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα. Από ό,τι φαίνεται σε άλλα κράτη και σε άλλες υπήρους ισχύει αυτό. Να λέμε, όποιος δεν τηρεί τους κανόνες και θα σας βοηθήσουμε βρε παιδιά να μάθετε τους κανόνες, ίσως και με ένα ενιαίο σύστημα πληροφορική, αλλά όποιος τηρεί τους κανόνες θα παίρνει τα κονδύλια. Όποιο δεν τους τηρεί, ε, δεν θα τα παίρνει. Τι να κάνουμε. Ε, πού είναι το πρόβλημα δεν καταλαβαίνω. Η στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει αυτή τη στιγμή και ε, το είπε και ο κύριος Λέβισον και χαίρομαι που το ελεγκτικό συνέδριο πάντα τα εξτάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια και σχολαστικότητα και είναι υπέρ του naming και shaming για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με γενικές διευθύνσεις και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί εδώ πέρα μας έχουν φέρει μια σαλάτα με στοιχεία και είναι λίγο περίπου σαν τη στρατηγική των Βρετανών στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τους βομβαρδίζανε με στοιχεία και πληροφορίες και δεν ξέρω ο αντίπαλος πού βρίσκεται. Λοιπόν, ε, να συνεργαστούμε με το ελεκτικό συνέδριο στην ανάλυση του ποιος ε, ε, εργάζεται καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιο λιγότερο. Υπάρχουν διαφορέ και από Γενική Διεύθυνση σε Γενική Διεύθυνση. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένω όμω να κατονομάζει και να διαπομπεύει και τα κράτη-μέλη. Naming and shame και εκεί. Όπω είπε και ο κύριο Μπαλσίτη, υπάρχουν ορισμένοι που παίζουν το παιχνίδι και δεν παίρνουν βοήθεια και άλλοι που δεν το παίζουν το παιχνίδι. Λοιπόν, να τα αναλύσουμε κάποια ώρα αυτά και για την κοινή γνώμη να έχουμε μια δομή που να την καταλαβαίνει και με διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη γιατί είχαμε και τη συνεδρία τη Επιτροπή ε, για την Περιφερειακή Ανάπτυξη ταυτόχρονα. Έπρεπε να παραστώ και στι δύο. Αλλά μετά πώς άκουσα σήμερα, ένα από τα κυρία στοιχεία είναι το εξή σημείο. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε το αμερικάνικο σύστημα και ρωτήσουμε τους Ευρωπαίους τι θα θέλανε να πάρουμε από το αμερικάνικο σύστημα ως προς την κεφάνεια, τελικά καταλήγουμε στο εξή. Μπορούμε να συγκρίνουμε συστήματα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν μόνο για την πολιτική συνοχή και βασίζονται στην μερισμένη η κοινή διαχείριση. Διότι η κοινή διαχείριση Ευρωπαϊκή Ένωση και 100 μελών και το πρόβλημα τη έλλειψη δεδομένων ή ελέγχου δεδομένων βασίζεται στην ευθύνη. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των συστηματών είναι ένα θέμα. Και η επιλεξιμότητα γνωρίζει δυσκολίε, όχι γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αναγκαστικά του κανόνε, αλλά γιατί διαφέρουν ευρωπαϊκοί από του εθνικού κανόνε και χάνεται ο κόσμο. Το θέμα είναι λοιπόν μπορούμε να έχουμε ένα σαφέ ευρωπαϊκό σύστημα του επιλέξιμου κόστου. Δεν υπάρχει ένα, ένα μοναδικό σύστημα δημοσίων προμηθειών. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν τους κανόνες οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί κανόνε από ένα κράτο στο άλλο όμω. Και δεν έχουμε πετύχει ένα ενιαίο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι δικό μα φάλμα. Πώ να συγκρίνουμε λοιπόν σύστημα ελέγχου και παρακολούθηση από του ίδιου του πολίτε, του κατοίκου, με το δικό μα. Εγώ διρωτώ με. Είναι συγκρίσιμα αυτά. Και ίσω οι Ευρωπαίοι οι ομιλητέ μα, αλλά και οι Αμερικανοί, είναι ενδιαφέρον να ακούσουν τη συζήτησή μα. Είναι το ίδιο αυτό που έχετε στις, Αμερικανικές, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την Ένωση, τα κράτη-μέλη και του δικαιούχου Και είναι πολύ περίπλοκη η διάδραση μεταξύ αυτών των ε, ε, επιπέδων. Υπάρχουν δημοσιονομικοί κανονισμοί και ούτω καθεξής. Τελικά θέλουμε να παρατήσουμε, να αφήσουμε κατά μέρο την κοινή διαχείριση, να την απλουστεύσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία. Εάν θέλει κανείς να υπερασπιστεί την κοινή διαχείριση ως επίτευγμα, πρέπει να παραδεχτεί ότι είναι πολύπλοκη από τη φύση της. Το θέμα είναι πόσο μακριά μπορούμε να πάμε σε αυτό το επίτευγμα. Ή θα την εκχωρήσουμε στα κράτη-μέλη, τα περισσότερα τουλάχιστον στοιχεία της κοινή διαχείρισης και θα είναι αυτά υπεύθυνα, ή θα αναρωτηθούμε αν θέλουμε να την διατηρήσουμε την κοινή και να την ελέγχουμε, να την παρακολουθούμε. Αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Δεν γίνονται όλα. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Πελεγκρίν, να προσθέσω και εγώ κάποιε παρατηρήσει. Είναι σίγουρα διαφορετικά τα πράγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση στι Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει από κεντρική πηγή ο έλεγχο για τα 800 ε, δολάρια, ενώ στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει πολλές ευθύνες εκ μέρου των κρατών μελών. Τώρα, για τα στοιχεία που μας δίνουν οι Ευρωπαϊκές Δυστικές Αρχές, η Όλαφ, τα άλλα ερευνητικά όργανα και ερευνητικά, ερευνητικοί οργανισμοί. Εντοπίζουν περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς και πολλές φορές εμπλέκονται και μέλη της κυβέρνησης των κατώμελών, των περιφερειακών κυβερνήσεων, εφόσον μιλάμε για ε, κονδύλια που διαχειρίζονται οι περιφέρειες, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή και σε εθνικό επίπεδο. Εκεί δεν ξέρουμε κατά πόσον οι ίδιοι έχουν ιδιαίτερο συμφέρον να παράσχουν τα στοιχεία και να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι επιπλέον λοιπόν προσπάθεια θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε σχέση με τα κάτι μέλη που δεν συνεργάζονται παρκώς με την, όλη αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τα ερχόμενα χρόνια βρίσκω. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Πελεγκρίν για να απαντήσει, μετά στην κυρία Μετερνόβα και μετά στον κύριο Λέβισον. Και στο τέλος, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε και εσείς ε, από την Αμερική, παρακαλώ. Ε, thank Um... Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Τι εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει ένα σύστημα αμερικανικού τύπου. Η απάντηση είναι ότι έχουμε τη συνυπευθυνότητα που κάνει τη διαφορά. Και ποια είναι η λύση να καταργήσουμε την από κοινού διαχείριση με τα κράτη-μέλη, δεν νομίζω αυτό να μπορούμε να το κάνουμε. Naming and shaming, να κατονομάζονται και να δημοσιεύονται αυτά, όχι μόνο για τα κράτη-μέλη και για τις γενικές διευθύνσεις. Θα μπορούσε να είναι Για τις κυρώσεις τώρα. Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο, αλλά μάλλον λιγότερο ρεαλιστικό στο παρόν πλαίσιο. Ο τρόπος που θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε είναι τα στοιχεία να είναι όσο γίνεται πιο χρήσιμα και πιο ακριβή. Και αυτό είναι καθήκον των κρατών μελών. Δεν ισχύει ότι μπορούν να παραμελήσουν να δίνουν ε, ακριβή στοιχεία τα κράτη-μέλη. Για, για τα χρήσιμα και τα ακριβή στοιχεία υπάρχει ελπίδα οι πολίτες και ε, να, να κάνουν κτήμα τους ε, αυτά τα στοιχεία και να πιέσουν τα κράτη-μέλη και τις ε, αρμόδιες αρχές να συμμετέχουν στη διαφάνεια και στην πρωτοβουλία αυτή. Uh, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα σχόλια για το τι θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ως δίδαγμα και τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον. Κατά πρώτον, αυτό που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο σχόλιο και ευνηδιάστηκα από έξω τα λόγια αυτά από μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, διότι αυτές ακριβώς οι συζητήσεις μας απασχόλησαν και στο διαλογό με τα κράτη-μέλη, είναι το εξής παράδειγμα. Το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιο ε, χρησιμοποιεί τα δημοσιοκομπήλια. Αυτό δεν είναι απλώ μια υπόθεση εργασία στην Εγγυρία Ήπειρο. Η προστασία δεδομένων και το πόρτο των επιχειρήσεων ήταν ακριβώς τα στοιχεία που μας απασχόλησαν από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΚΟΚΟΦ ε, ετοιμάσαμε τι κατευθυντηρίε γραμμέ μα για δημοσίευση προ του δικαιούχου. Και ε, το σχόλιο που ε, λαμβάναμε ήταν ε, για ποια εμπιστευτική πληροφορία των εταιριών μιλάμε. μιλάμε για δημόσια κονδύλια. Το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει. Πιστέψτε με, από τα μέλη που προσχώρησαν το 2004 και το 2007, τις αντιρρήσεις δεν τις προέβαλαν αυτές οι χώρες, οι καινούργιες. Αλλά τα δυσκολίε τι είχαμε με τι χώρε που ήταν πολλά χρόνια νωρίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούσαν τι ε, συνεισφορέ των διευθυντικών ταμείων, τι γεωργικέ επιδοτήσει ε, πολλά χρόνια, όχι με την αντιπροεδρία της Εστονία το 2005. Έτσι λοιπόν, με το έγγραφό μα, με τι κατευθυντήριε γραμμέ και τη σχετική συζήτηση, το βασικό θέμα ήταν η προστασία των δεδομένων, ε, η εμπιστευτικότητα των ε, επιχειρηματικών πληροφοριών και από τη δική μου πλευρά και σε ό,τι αφορά τι περιφέρειε, μπορώ να σα διασφαλίσω ότι κανένα πρόβλημα δεν θα είχα να διαπομπεύω του ε, υπευθύνου των γενικών διευθύνσεων του Name and Shame. Εδώ πραγματικά τα κράτη-μέλη μείναν στο ελάχιστο επίπεδο που θέλαμε να διασφαλίσουμε και βάσει της ε, αποκοινό διαχείρισης που θέλουμε να πετύχουμε και που διαθέτουμε για αυτόν τον περίοδο προγραμματισμού έχουμε πιέσει τα πράγματα όσο περισσότερο γινόταν. Και έχουμε και το επαναλαμβάνω το παράδειγμα της Λιθουανίας είναι εξαιρετικό και το Ουγγρικό είναι πολύ καλό. Οι χώρες τα πήγαν πολύ καλά. Ξεπέρασαν μάλιστα το όσα όριζαν οι κανόνες και Για, στο δικό μας μυαλό ο κατάλογος των δικαιούχων στόχο δεν είχε να κάνει διασταυρούμενε συγκρίσει και διασταυρώσει δεδομένων μεταξύ κρατών μελών. Αυτό που θέλαμε να πετύχουμε είναι ο το κοινό στα κράτη-μέλη, οι πολίτε να έχουν δυνατότητα να γνωρίζουν. Γιατί έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν. Δυνατότητα ε, ε, ε, διερεύνηση λοιπόν και ένα σύστημα φιλικό προς το χρήστη. Όχι θεωρητική σύγκριση και συλλογή δεδομένων και δυνατότητα έρευνας. Δεν ήταν ε, θεωρητική η αναζήτησή μας. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι την ευκαιρία την επόμενη φορά θα πρέπει να την αντράξουμε όταν ε, νομοθετικώς θα πρέπει να αποφασίσουμε για το επερχόμενο διάστημα προγραμματισμού. Ξέρετε ότι η Επιτροπή έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας και για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία που ήρθε το 2005, ξέρετε ότι οι κανονισμοί είχαν συνταχθεί νωρίτερα. Δεν είχαμε το χρόνο ίσως να τα σκεφτούμε όσο έπρεπε και του χρόνου θα αλλάξουν τα πράγματα όταν θα ετοιμάσουμε τα κείμενα για το ερχόμενο διάστημα προγραμματισμού. Όμως η διαδικασία διαπραγματεύσεων, ό,τι και αν τελικά αποφασίσει η Επιτροπή, θα πρέπει να γίνει και στο Συμβούλιο και οι μαγικές ε, συνταγές, τα μαγικά αυτά λόγια και οι φόρμουλες για την εμπιστευτικότητα των στοιχείων των εταιριών και την ε, προστασία των δεδομένων σίγουρα θα ανακύψουν και πάλι γιατί οι πολιτιστικές προτιμήσεις, οι πολιτικές ε, προτιμήσεις των κρατομελών σίγουρα έρχονται εδώ να επηρεάσουν το σκηνικό όταν μιλούμε για τέτοια θέματα. Διαφέρουν αυτά από την, το σύστημα οικονομική ανάκτηση, όπως το διαχειρίζεται κεντρικό η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όμω, πράγματι, νομίζω και θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο Πευσιών ότι η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Τα ζητήματα λοιπόν της προστασίας προστασία των δεδομένων και τη εμπιστευτικότητα των εταιρικών στοιχείων δεν έχουν εδώ καμία σχέση. Και να είναι ενήμεροι οι μελλοντικοί δικαιούχοι είναι σημαντικό και η δημοσίευση του καταλόγου των δικαιούχων εξίσου. Και αυτό αφορά το σύνολο του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού κατά τη δική μας άποψη, όχι μόνο την πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λέβισον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας είχα πει ήδη ότι το συνέδριο δεν θα μπορέσει να σας κάνει πολιτικές δηλώσεις εδώ. Αλλά θα σας πω τι νομίζω ότι θα κάνουν οι διάδοχοί μας το 25 όταν θα κάνουν την αποτίμηση αυτής της πρωτοβουλίας. Αν είχατε ακούσει αυτά που σας είπα θα καταλάβατε ότι άκουσα την κυρία Πελεγκρίν, ίσως να την παρεξήγησα, αλλά δεν νομίζω ότι μέχρι τώρα υπήρξε κανένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης της διαφανείας. Το 25 λέμε ότι καλό θα ήταν είχε υπάρξει, να είχε υπάρξει συμφωνία μέχρι τότε μεταξύ των ενδιαφερομένων. Γιατί εδώ βλέπουμε στρατηγούς να προπορεύονται του στρατού κατά 25 μίλια. Και η οπισθοφυλακή τι θα γίνει. Εδώ τα μέλη της Κοκομπούς ενδιαφέρονται περισσότερο από ότι οι πολίτες και οι επιχειρηματίες. Άρα καλό θα ήταν να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη συνοχή για να το πω έτσι και σε αυτά τα θέματα. Οι στόχοι του SMART τώρα εννοούν όπως σας είπα τον κατάλογο των αρχικών που είχα αναφέρει λοιπόν. Αλλά και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων ελπίζω οι διάδοχοι μου το 2025 να το καταλάβουν. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Με χαρά όμως βλέπω, ακούω uh, ότι τουλάχιστον οι στόχοι έχουν διατυπωθεί προς το κοινό, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ντέβενη, κύριε Μπρίτο, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ε, για μένα ήταν συναρπαστικό να ακούσω τη σημερινή συζήτηση. Τη συζήτηση που είχατε μεταξύ σα. Μου θυμίζει τη συζήτηση που άκουζα, άκουγα ε, πριν από δύο χρόνια σχετικά με τα θέματα αυτά στι ΗΠΑ. Και Σήμερα έχουμε καταλήξει σε ένα κεντρικό σύστημα, αλλά αυτό δεν έγινε εύκολα. Πολλά από τα ζητήματα που ανέκυψαν και εδώ, ζητήματα ειδικού βίου, προστασία δεδομένων, απροθυμία παροχή δεδομένων, όλα αυτά. Και, ε, και τους Αμερικανούς ε, γερουσιαστές απασχόλησαν. Επίσης υπήρξαν ε, πολλές ομάδες ε, πίεσης υπέρ της διαφάνειας που πίεζαν για μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες. Τώρα, το σύστημα που διαχειριζόμαστε τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν είναι η πρώτη προσπάθεια να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είχαμε και άλλα συστήματα την τελευταία δεκαετία και το καθένα τους είχε κάποια σχετική επιτυχία και κάποια, μπορούμε να πούμε, και κάποια αποτυχία. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος και αυτό ήταν μεγάλο όφελος για να φτιάξουμε το σημερινό σύστημα. Μου έκανε εντύπωση που τέθηκαν τα εξή ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα τι πρέπει να συλλέγεται, τι δεδομένα πρέπει να συλλέγονται. Αυτό μου αυτό μου κάνει να σκεφτώ ότι με του κανόνε που θα πρέπει να συντάξετε και να προβλέψετε στο μέλλον θα μπορείτε να το λύσετε αυτό. Μετά πώ θα γίνεται η συλλογή. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Εγώ σα εξήγησα ότι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα για τη συλλογή δεδομένων, διότι ειλικρινώ όλοι οι ομοσπονδιακοί φορεί και οργανισμοί έχουν συστήματα, αλλά ξεχωριστά. Σε διαφορετική κατάσταση ετοιμότητα το καθένα. Και το Τρίτο θέμα είναι πώς θέλουμε να εμφανίζονται, να δημοσιεύονται τα στοιχεία. Εάν θα είναι ένα ιστότοπος ανοιχτό σε όλους, διδραστικός, που θα περιέχει στοιχεία που δεν προϋπήρχαν ποτέ σε κυβερνητικό ιστότοπο. Ίσως να σας ακούγεται ότι είμαστε κάπως πιο προχωρημένοι, γιατί έχουμε ένα σύστημα λιγότερο αποκεντρωμένο. Αλλά να σας πω τη δική μου άποψη, αν δεν είχε μεσολαβήσει η οικονομική κρίση, δεν θα είχαμε τέτοιο σύστημα σήμερα, πιστεύω. Οι προσπάθειες λοιπόν για ένα κεντρικό σύστημα στην Ευρώπη σίγουρα έχουν να κάνουν και με την ιδέα ότι πολίτες έχουν δικαίωμα να μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία αυτά. Το κάνουν, δεν το κάνουν. Αυτό το ακούσαμε πολλές φορές σήμερα και το βρίσκω σωστό. Ευχαριστώ. Να πω προς το απόρριτο και την προστασία των δεδομένων από τη δική μας πείρα στις ΗΠΑ δεν ήταν ότι δεν είχαμε καμία επιλογή. Αλλά δεν μπορούσαμε να πούμε και η άσπρη μαύρο, δηλαδή όλα τα στοιχεία να εμφανίζονται ή όχι. Ε, για τις επιχειρήσεις που απευθείας έχουν ε, συναλλαγές με την κυβέρνηση, κάποιοι διαγωνισμοί ε, βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια και μπορεί να επηρεάζουν και άλλες εταιρείες. Λοιπόν, ο τομέας αυτός μπορεί να μην ε, εμφανίζεται δημοσίως, αλλά το τι σύμβαση πήρε μια επιχείρηση, γιατί πόσο, με, ποια, με ποιο σκοπό, αυτά συνήθως δημοσιοποιούνται. Και το θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές φορές ήταν ιδιωτικό βίος, σας είπα νωρίτερα, για τους φόρους, πώς οι τοπικές κυβερνήσεις απαιτούν Ε, οι τοπικές αρχές να λογοδοτούν σε επίπεδο σχολείων για το τι ξοδεύουν πού, για τους δασκάλους λόγου χάρη. Ο καθένας θα μπορούσε να συλλέγει δεδομένα για την αμοιβή, το μισθό του κάθε δασκάλου και το τι ακριβώ κάνει. Ίσως αυτό θα ήταν μια καλή ιδέα, αλλά για την ώρα δεν γίνεται. Ξέρουμε απλώ τον αριθμό των δασκάλων, έχουμε ένα μέσο όρο για του δασκάλου, για εργαζομένου στα σχολεία, κάπω έτσι. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί κανεί ε, ω προ την προστασία των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα να τα καλύψει τα ζητήματα αυτά, χωρί να τα βλέπει απόλυτα και να ικανοποιεί και του στόχου τη διαφάνεια. Πρόεδρο, ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Γκρέσλε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θυμίσω στην ερώτησή μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία ε, Πελεγκρίνη. Ποια είναι τα κράτη-μέλη και ποιες οι περιφέρειες που έχουν πολύ κακές επιδόσεις τα γνωρίζουμε αυτά. Έχουμε επίγνωση και ποιοι έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Έχουμε ένα ranking έτσι με 27. Για κατάταξη, εν περιπτώσει, να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Μέχρι σήμερα ε, αυτή η υποχρεωτική δήλωση ε, απέτυχε. Είχε καλές προθέσεις, αλλά κακή υλοποίηση. Και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την επιτυχία γιατί έχει ε, εφαρμοστεί πάρα πολύ άσχημα. Ερωτώ τώρα το ελεκτικό συνέδριο. Πότε ε, έχετε προγραμματίσει τον επόμενο έλεγχο. Κάτι άκουσα 2025, αλλά νομίζω ότι με ε, απατούν τα αυτιά μου. Δεν φαντάζομαι μέχρι το 2025 να περιμένετε. Και αν θέλετε να υπάρξει ένα στοιχειώδης κοινοβουλευτικός Έλεγχο, τότε πάρτε καμιά φιλιά να κρεμαστείτε. Γιατί τι να ελέγξουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Τι γίνεται με τι διοικητικέ δαπάνε, τι μα δίνει από ενημέρωση το ελεκτικό συνέδριο για να ξέρουμε ποια προγράμματα την χάνουν και ποια όχι. Ζήτησα διοικητικέ δαπάνε και ακούω κάτι πράγματα εξωφρενικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι γνωρίζουμε για τι διοικητικέ δαπάνε, τι γνωρίζουμε για την επιτυχία τέτοιων πρωτοβολιών, γιατί τώρα θα πρέπει να κάνουμε την ε, τελική ρύθμιση. Και κάτι άλλο, ω εισηγήτρια για το δημοσιονομικό κανονισμό, μαθαίνω συνεχώ, γιατί είναι και τριετή αυτή η προσπάθεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα κεντρικό σύστημα με σαφή στοιχεία. Ποια ε, δεδομένα βάζουμε στο σύστημα σε μία γλώσσα, σε ένα νόμισμα και μία φορά το χρόνο αξιολόγηση αρχίζει γενομένη από αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή ποιο παίρνει τα λεφτά και τι τα κάνει. Με έναν τρόπο δομημένο, καθαρό, ε, ξέρουμε τι γίνεται. Και κύριε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σας πω το συναρπαστικό που ακούσαμε, αυτό που είπατε κύριε Ντέβεν στην αρχή, 50 υπάλληλοι ε, στη Washington και 329 επιθεωρητές και έχετε 8.000 στην Ευρώπη υπαλλήλους. Αν τους προσθέσω όλους, μάλλον αυτό συνολικά στις ΗΠΑ, για, ε, για πολύ λιγότερα χρήματα. Εμάς είναι 125 δισεκατομμύρια το χρόνο. 125 δις. Και πόσα λίγα μας δίνουν αυτοί που δουλεύουν εκεί. Και να θεωρεί και το ελεκτικό συνέδριο ότι τον αφορούν αυτά που, λέω. Δεν σας κοιτάω τυχαία, ούτε έτσι αθώα. Αυτά. Grazie, onorevole Andreas. Ευχαριστούμε κυρία Ανδρέας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ανέφερε η κυρία Πελεγκρίν την Ισπανία και την Πολωνία και είπε ότι είναι απρόθυμε να δημοσιεύσουν πληροφορίε για του δικαιούχου του. Εγώ ρωτώ την Επιτροπή, τι μέτρα ελήφθησαν ώστε η Πολωνία και η Ισπανία να αποχρεωθούν να δημοσιεύσουν τι πληροφορίε. Και επίση ρωτώ την Επιτροπή, γιατί να μην γίνει κριτήριο για την ε, επιστροφή ή διαφάνεια, ο σεβασμό τη διαφάνεια. Ευχαριστούμε, κυρία Πελεγκρίν, για να απαντήσει στην κυρία Γκρέσλε. σε ό,τι αφορά τον καθορισμό καταλόγου καλών επιδόσεων και κακών επιδόσεων, καλών και κακών μαθητών, δεν μπορώ να πω ότι έχω διεξοδικό κατάλογο, οπότε αισθάνομαι κάπω άβολα και το να κατονομάσω συγκεκριμένε περιπτώσει δεν θα ήταν πολύ δίκαιο όμω. Πρώτη στον κατάλογο είναι η Φιλανδία και η Γαλλία και τελευταίοι θα ήταν η Ιταλία. Μάλλον, σε ορισμένε τουλάχιστον περιφερειέ τη. Η Ισπανία νομίζω έχει βελτιωθεί πολύ. Συγγνώμη που είναι έτσι άδικη η επίδειξη στοιχείων, αλλά... Ευχαριστούμε για αυτές τις πληροφορίες. Για μένα δεν είναι καινούρια τα νέα, σε ό,τι αφορά την Ιταλία, κύριε Ματερνόβα. Ευχαριστώ. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω λίγο να ταξινομήσω τα πράγματα δεν έχουμε πλήρη συγκρί, πλήρως συγκρίσιμα στοιχεία, ούτε το στοχεύσαμε άλλωστε ποτέ. Αλλά να σας ενημερώσω από αυτόν που είπε η κυρία Πελεγκρίν, μας ανέφερε τις γκρίζες ζώνες του χάρτη. Δεν είναι πια γκρίζες αυτές οι ζώνες τώρα. Όλες οι χώρες έχουν συμμορφωθεί. Η Ισπανία ήταν από τις τελευταίες αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι το σύστημά της δεν είναι αξιόπιστο. Η Ισπανία, η Ελλάδα, μερικές περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου και η Ιταλία ήταν οι τελευταίες. Το ισπανικό σύστημα πάντως δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Όπως είχε πει η κυρία Πελεγκρίν για το Ιταλικό δηλαδή. Με την Πολωνία δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα εδώ νομίζω υπήρξε παρεξήγηση. Η Πολωνία ποτέ για μας δεν υπήρξε πρόβλημα ως προς τη δημοσίευση των ωφελουμένων. Γενικά, η εμπειρία μας λέει ότι όσο πιο αποκεντρωμένο είναι ένα κράτος, τόσο πιο, δύσκολο, πιο δύσκολη η δημοσίευση των στοιχείων του στις ομοσπονδιακές χώρες αυτό πάντα υπήρξε πρόβλημα. Οι νέες χώρες ήλπιζαν, κατά τραγική ηρωνία, ότι η δημοσίευση συμβαδίζει με τη χορήγηση των χρημάτων, αλλά... Τελικά, με τις καινούργιες χώρες συνεννοηθήκαμε πιο εύκολα. Παραδείγματος χάρη η Λιθουανία και η Ουγγαρία είναι από τις καλύτερες μας περιπτώσεις. Ενώ η Δανία, η Σουηδία και η Φιλανδία και αυτές, και αυτές έχουν πολύ καλές ιστοσελίδες, πολύ καλές. Και δεν έχω άλλες πληροφορίες για μεμονωμένες χώρες μέλη. Για τα σχόλια της κυρίας Γκρέσλε για ενιαίο νόμισμα, ενιαία γλώσσα, ενιαίο σύστημα. Το κατά πόσον είναι ευκταία η χορήγηση των πληροφοριών, είναι και πολιτικό θέμα και δεν είμαι βέβαιη ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μας ανέθεταν ποτέ θα μας έδιναν ποτέ τη δικαιοδοσία που θα σήμαιναν αυτά που ζήτησε η κυρία Γκρέσλε. Η Επιτροπή γνωρίζει ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της στις διαθεσμικές σχέσεις δεν κάναμε καν τη σχετική πρόταση γιατί προσπαθούμε να είμαστε υπεύθυνοι και ρεαλιστέ και ρεαλίστριες ως προς το τι είναι νομοθετικά δυνατόν. Επαναλαμβάνω όμως ότι μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο αυτά που καταφέραμε είναι ουσιώδη και ένας από τους αξιοτήμους κυρίους βουλευτάς είπε προηγουμένως ότι δεν έχει προβλεφθεί καμία στήριξη του συστήματος για τις χώρες. Αλλά πώς έχουμε οργανώσει σεμινάρια, πράγματα και, και αυτός είναι ένας τρόπος να τους βοηθήσουμε για να μεταφερθεί η γνώση αυτή και αλλού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Λέβισον. Ευχαριστώ. Άκουσα τα ερωτήματα της κυρίας Γκρέσλε και ελπίζω να μην ακούστηκε ειρωνικός όταν μίλησα για το 2025. Απλώς σκεφτόμουν ότι απαραίτητο είναι να το σκεφτούμε από τώρα. Πρέπει να εξεύρουμε κάποια στρατηγική. Να δούμε ποιος είναι ο στόχος του συστήματος που θέλουμε να σχεδιάσουμε να βελτιωθεί το σύστημα που σχετίζεται με αυτή την πρωτοβουλία. Γι' αυτό πρότεινα να χρησιμοποιούμε τους στόχους SMART, αυτούς τους ευθύς στόχους. Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Ίσως όχι στο τόσο απότερο μέλλον, ίσως ήδη στο 2014 να μπορούμε στο ελεγκτικό συνέδριο κάτι να κάνουμε για όλα αυτά. Όμως, προτού γίνει κάτι σε επίπεδο, θα χρειαστούν και πολιτικές πρωτοβουλίες. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν νομίζω ότι μπορεί να επιληφθεί μόνο του του θέματος. Διότι όπως άκουσα και τώρα από την κυρία Πελεγκρίν, εάν εμείς επιληφθούμε, δεν θα έχουμε και πολλά να κάνουμε. Δεν θα βελτιώσουμε λοιπόν ούτε τα δικά της τα πορίσματα σε αυτή τη φάση. Δεν θα υπάρχει αντικείμενο εάν ξεκινήσουμε από το 2010 και προσπαθήσουμε να συντάξουμε μια έκθεση. Θα έλεγα λοιπόν να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις πρώτα και να βασιστούν και στην απλούστευση και να λάβετε υπόψη την ε, ιδιαίτερη φύση αυτής της περιοχής. Όταν ε, δεν ξέρω αν συνηθίζεται να μιλάμε για συγκεκριμένε περιπτώσεις. Ας πούμε ότι χτίζουμε μια γέφυρα μεταξύ Δανίας και Σουηδία. και ε, μπορεί να μπουν δύο ονόματα στον κατάλογο στα στοιχεία, αλλά να εμπλέκονται εδώ εκατομμύρια ευρώ και να είναι δεκάδες οι συνεργάτες. Στο χτίσιμο λοιπόν μιας γέφυρας μπορεί να προκύψουν και πολλές περιπτώσεις δικαστικές. Άρα το ζήτημα είναι να σκεφτούμε και τι θέλουμε να δημοσιεύουμε ένα τομέα. Για μένα αυτό είναι καθοριστική σημασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπαλτσίτης έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα αναφέρθηκε ότι εδώ συζητούμε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Συμφωνώ με αυτό. Τη μία την παρουσίασαν οι επισκέπτες μας, και βασίζεται στο τι επικρατούσε και συζητιόταν πριν από 10 για 15 χρόνια και η άλλη βασίζεται στην τάση να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα. Σωστά το είπε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Συνεδρίου. Πρέπει να λάβουμε πολιτικές αποφάσεις στο μέλλον. Πρέπει να ληφθούν και ίσως τότε θα έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Ίσως λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ξανασκεφτεί τα ζητήματα αυτά και στο μέλλον. Αλλά έως τότε οι επισκέπτες μας θα μπορούσαν ενδεχομένω να μα δώσουν τουλάχιστον τα αριθμητικά, στοιχεία για το προσωπικό και το πώ θα μπορούσε το προσωπικό αυτό να επιδιώξει του στόχου και βάσει συγκεκριμένων προτάσεων να αποφασίσουμε για το μέλλον. Διότι είδαμε ότι η συνεργασία μεταξύ γενικών διευθύνσεων δεν έχει πετύχει ως τώρα επαρκώς. Οπότε α ακούσουμε τις απόψει των επισκεπτών μας και του κυρίου Λιμπεράτσικη που παρουσίασε την όλη ακρόαση. Ναι, θα δώσω το λόγο για τις απαντήσει και μετά στον κύριο Λιμπεράτσικη για το συμπέρασμα. Κάποιο θα ήθελε να σχολιάσει, τόσο από ο κύριο Μπαρτσίτη, Η Επιτροπή ίσως. Όχι. Ο κύριος Λιμπεράτσικη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχει περάσει ο χρόνος μας, γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πρώτον, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι είναι κοινό και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνονται σφάλματα και απάτες. Άρα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε φαντάζομαι. Δεύτερη παρατήρηση. Τι έμαθα από εσά σήμερα κύριε Τεβάνη. Ναι η ιδιωτική σφαίρα είναι οι πόροι. Όταν χρησιμοποιείς δημόσιους πόρους είναι άλλα δημόσια. Δεν υπάρχει προστασία ιδιωτική ζωής. Αυτά λέει η αμερικανική προσέγγιση. Εμείς έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για την ιδιωτική σφαίρα. Ε, στη συνέχεια η διαφάνεια δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ένα εργαλείο, λέει ο κύριος Βρήτο. Άρα είναι ένα εργαλείο για να γίνεται χρηστή διαχείριση των πόρων. Τέταρτον, Περισσότερη διαφάνεια, καλύτερη ένωση. Αυτά μας λέει το ελεγκτικό συνέδριο και ο κύριος Λέβισον. Και ε, το ελεγκτικό συνέδριο εκπροσωπείται εδώ κατά το 1 του 5 έχουν έρθει πολλά μέλη. Πέμπτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να είναι υπεύθυνη για καλύτερη ένωση. Ας θυμίσουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι επίσης μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να φοβάται ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη-μέλη. Εμείς δίνουμε την απαλλαγή εδώ πέρα, η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο. Ε, και Κύριε Πρόεδρε Ματζίστρη, σας ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη σας να δώσετε ευκαιρία να γίνει αυτή η ακρόαση. Ευχαριστώ όλους όσοι συνεισέφεραν και όλους εκείνους που έλαβαν το λόγο, καθώς επίσης και το κοινό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για το δικό σας έργο. Ευχαριστώ και τους επισκέπτες μας. Ευχαριστώ τους δύο Αμερικανούς φίλους. Πραγματικά η συνεισφορά τους ήταν πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ για την όλη συζήτηση. Θα σας δούμε την επόμενη φορά. Αντίο σας.